<laughs> Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ καθίστε. Γιατί κανονικά ήδη έπρεπε εδώ και 10 λεπτά να είχαμε ξεκινήσει τη συνεδρίασή μα. Στην ημερήσια διάταξη, στο σημείο 11, το σχέδιο έκθεση τη κυρία Μακιντάιρ θα συζητηθεί αύριο μετά το 22. Και όχι στη θέση του στο 11 δηλαδή. Και το σημείο 18 η ψηφοφορία για την ε, γνωμοδότηση του κυρίου Χόουιτ αναβάλλεται για τις 9 Δεκεμβρίου. Θα συζητήσουμε σήμερα την γραμματότηση Χόουιτ, αλλά δεν θα ψηφίσουμε αύριο. Υπάρχουν σχόλια για την ημέρηση διάταξη. Όχι, οπότε τροποποιείται όπως σας προανέφερα. Τώρα, σημείο 2. Ανακοινώσεις της Προέδρου. Έξι ανακοινώσεις έχω. Πρώτον, σε ό,τι αφορά το εργαστήριο για την, την οργάνωση που φορά την α, ασφαλέστερη εργασία σε κάθε ηλικία. Θα γίνει τη Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 3.30 με 6.30 και σας προσκαλώ στην διοργάνωση αυτού του εργαστήριου. Ελάτε παρακαλώ όσοι μπορείτε. Ε, ζητώ συγγνώμη που περνάω τη μια γλώσσα στην άλλη από του διερμηνεί, γιατί ξέρω ότι του ενοχλεί αλλά μερικέ φορέ έχω μπροστά μου το έγγραφο στα αγγλικά και είναι πιο εύκολο. Λοιπόν, δεύτερο θέμα ε, ε, συνεδρίαση τη 9 η Ιανουαρίου του 2014. Παρακαλώ, σημειώστε το. Σα το είχα προαναγγείλει και στην προηγούμενη έκτακτη συνεδρίαση που είχαμε στο Στρασβούργο επαναλαμβάνω, 5η 9 Ιανουαρίου 2014 το πρωί. Τρίτη ανακοίνωση. Ευρωπαϊκή Κοινοβουλευτική Εβδομάδα για το 2014. Τότε που συζητούμε με τα Εθνικά Κοινοβούλια για θέματα που αφορούν το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και την εφαρμογή του άρθρου 13. Διακόπτη πρόεδρος. Αυτή η Ευρωπαϊκή Κοινοβουλευτική Εβδομάδα αφορά και το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και τη διάσκεψη που προβλέπει το άρθρο 13 της συνθήκης για τη σταθερότητα, το συντονισμό και τη διακυβέρνηση στην ε, Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Αυτή η εβδομάδα θα γίνει φέτος 20 με 22 Ιανουαρίου 2014. Θα σας στείλουμε σύντομα τις, επο... τις ε, συγκεκριμένες ε, ημερομιές και πρόγραμμα. Περιμένουμε τις προτάσεις της Ελλάδας ε, για τις ε, αρμοδιότητες των διαφόρων ε, συνεδριάσεων που προβλέπει το άρθρο 13. Επίσης, θα έχουμε διακοινοβουλευτική συνεδρίαση των Επιτροπών με δύο θέματα. Καταρχήν, την κοινωνική διάσταση της ΟΝΕ, της Οικονομικής και Νομισματικής Επιτροπής και Ένωσης και δεύτερον, τα θέματα της αιτήσιας επισκόπης για την ανάπτυξη, κυρίως εγγύηση των νέων, μεταρρύθμιση των συντάξεων και η ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Αυτά τα θέματα θα συμπεριληφθούν σε ένα κοινό κεφάλαιο που ανταποκρίνεται στην εξέταση της ετήσιας επισκόπησης για την ανάπτυξη σε συντονισμό που έγινε προηγουμένως με συντονιστές και μάλιστα δύο φορές. Αυτή η διακοινοβουλευτική συνεδρίαση θα γίνει την Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 9 με 11.30 οπότε παρακαλώ σημειώστε το ήδη από τώρα για να έρθετε στην συνάντηση αυτή όσο πιο πολύ γίνεται. Σημείο 4. Ανακοίνωση 4. Είχαμε συμφωνήσει με τους συντονιστές ε, στην τελευταία συνεδρία των συντονιστών να δημοσιεύσουμε μετά την συνεδρίαση που είχαμε με τον Επίτροπο Άντορ για την εφαρμογή των συμφωνιών των κοινωνικών εταίρων. Συμφωνήσαμε λοιπόν να δημοσιεύσουμε μία ανακοίνωση τύπου. Τη μοιράσαμε στους συντονιστές και τρεις κοινοβουλευτικές ομάδες ήδη αντιτάχθηκαν στη δημοσίευση της, αυτού του ανακοινωθέντος τύπου. Κάτι που ερχόταν σε αντίθεση με την ήδη λυμμένη απόφαση των συντονιστών. Προτείνω λοιπόν μέχρι το βράδυ να θεσπίσουμε μία προθεσμία υποβολής τροπολογιών ώστε να μπορέσουν όλοι να υποβάλουν προτάσεις αντί απλώς να απορρίπτουν ε, την πρόταση των συντονιστών ε, που ήδη είχαν αποφασίσει για τη δημοσίευση των ανακοινοθέντων τύπου. Θα σας ε, υποβάλω αργότερα μία σύνοψη πρότασης που θα υποβάλω και αύριο στους ε, συντονιστές προς έγκριση. Ανακοίνωση 5. Δεν είχαμε διερμηνία χρησιμοποιητή. Α, συγγνώμη. Είχαμε διερμηνία που δεν χρησιμοποιήθηκε. Α, μεταξύ γαλλικών και αγγλικών για την έκθεση Howitt σε μια συνεδρίαση που έγινε με τους κοιόδης ηγητές. Εκεί ο κύριος Μπουλόν, παρόλο που είχε ζητήσει διερμηνία, απουσίασε και έτσι δεν χρειάστηκε διερμηνία προς τα γαλλικά πολλές από αυτές τις πληροφορίες αφορούν το ΕΛΚΑ που έχει μόνο ένα μέλλον παρόν και κανέναν να βοηθώ. Ελπίζω να διαμηνυθούν όλα αυτά τα στοιχεία στο ΕΛΚΑ. Επίσης τα πρακτικά μοιράστηκαν ηλεκτρονικά και ε, υπάρχει και η όλη τεκμηρίωση στην, στον ιστότοπό μας, στον ιστότοπο της Επιτροπής μας. Σας παραπέμπω εκεί. Αυτές ήταν λοιπόν οι έξι ανακοινώσεις της Πρόεδρου και μπορούμε να περάσουμε στο σημείο 3 που προβλέπει εξέταση των τροπολογιών της γνωμοδότησης του κ. Χόουιτ. Θα εξετάσουμε ταυτόχρονα και τις τροπολογίες και τις συμβαστικές τροπολογίες. Τέσσερις είναι οι συμβαστικές τροπολογίες. Ε, ο κύριος Χόουιτ θα συντάξει γνωμοδότηση που θα επιδώσει στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων με θέμα τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυμορφία από ορισμένε μεγάλε εταιρείε και ομίλου. Κύριε Χόουιτ, έχετε το λόγο. Thank you very much indeed. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Να θυμίσω σε όλους εν είδη εισαγωγής ότι είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η οδηγία που προωθεί ο Επίτροπος Μπαγνιέ και χέρι ευρείας υποστήριξης από όλους, ιδίως μεταξύ της επιχειρηματικής κοινότητας πάρα πολλές επιχειρήσεις συμμετέχουν στην πρωτοβουλία ε, για την ε, σύνταξη κοινωνικών απολογισμών. Περίπου χίλιες εταιρείες ε, οι οποίες εκδίδουν απολογισμούς για τη βιώσιμη ανάπτυξη και προσπαθούν για να τεκμηριώσουν και τις προσπάθειές τους για ένα πιο αηφόρο οικονομικό μέλλον. Όλες αυτές οι εταιρείες, επί της αρχής τουλάχιστον, είναι υπέρ αυτής της νομοθεσίας. Ε, είναι μια κεντροδεξιά επιτροπή, όχι μια κεντροαριστερή επιτροπή αυτή της οποίας προείσταται ο κύριος Μπαρνιέ. Και όπως είπα πολλές, όπως πολλές φορές έχει συμβεί εδώ στην Επιτροπή μας, ε, έχει τεθεί το θέμα για την υιοθέτηση νομοθεσίας, αλλά πάντοτε υπήρχαν αντιρρήσεις. Και πέρυσι το κάναμε με συμβιβαστικές προτάσεις ε, μεταξύ της του ΕΛΚ και άλλων πολιτικών ομάδων και ελπίζω να περάσει αυτή τη φορά. Επίσης πιστεύω ότι το να έχει κανείς ενοποιημένους ε, νομοθεσμία και τους ενοποιημένους απολογισμούς και όχι να ε, θεσπίζονται πρόσθετες υποχρεώσεις για τις επιχειρήσεις είναι θεμελιώδους ε, σημασίας. Να αντικατοπτρίζονται όλα αυτά τα στοιχεία στους ετήσιους ε, οικονομικούς απολογισμούς που ούτως ή άλλως συντάσσουν οι εταιρείες. Υπάρχουν όμως θέματα κατά πόσο η Επιτροπή θα πρέπει να εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές. Εγώ το είμαι υπέρ. Εάν θα πρέπει να πούμε λίγα πιο ξεκάθαρα τα πράγματα τα σχετικά με την επιβολή του νόμου, αν και το μεγαλύτερο μέρος της αρμοδιότητας θα ανήκει στα κράτη-μέλη. Ε, σήμερα το απόγευμα στην συζήτηση μπορούμε να συζητήσουμε όλους τους συμβιβασμούς. Εκεί που προσπάθησα να επιτύχω συμβιβασμού σε δύο συναντήσεις την προηγούμενη εβδομάδα και έχω σημειώσει πρόοδο, είχα και ξεχωριστή συνάντηση με τον Σκιώδη ε, εισηγητή από το ΕΛΚ τελικά συναντηθήκαμε χθε το βράδυ, έκανε τη διερμηνέα η γραμματέας μου και μπορώ να πω ότι σημειώσαμε αρκετή πρόοδο και τον ευχαριστώ. Λοιπόν, για τις συμβιβαστικές προτάσεις προσπάθησα πρώτον να μείνουμε όσο το δυνατόν πιο κοντά στις προτάσεις του κυρίου Μπαγνιέ. Να μην προσπαθήσουμε να κινηθούμε εμεί προς άλλη κατεύθυνση ως το κοινολούγιο. Εγώ ήμουν προετοιμασμένο, κοιτάζοντας τις τροπολογίες του ΕΛΚ, να επιλέξω μερικά πράγματα ε, τα οποία πάνε προς τη σωστή κατεύθυνση και ε, η προσθήκη για παράδειγμα της φράσης where relevant, όπου αρμόζει, ε, και επίσης η όλη φρασεολογία για το ουσιώδες, για το materiality, έχω και την στήριξη του κυρίου Μπίλονγκ και στηρίζω τις τροπολογίες του και τις κοινωνικές επενδύσεις. Ε, διατηρώ μια επεξηγηματική και διευκρινιστική προσέγγιση. Πιστεύω ότι υπάρχει μια παρεξήγηση εδώ. Ή ο κόσμος των επιχειρήσεων μας ζητά να έχουμε μια τέτοια προσέγγιση, μια μία προσέγγιση συμμόρφωσης. Νομίζω ότι η Επιτροπή προσπαθεί να σκληρύνει την νομοθεσία για τις επιχειρήσεις. Αυτή η προσέγγιση comply or explain, δηλαδή θα συμμορφωθείς ή θα εξηγήσεις τους λόγους για τους οποίους δεν συμμορφώνεσαι, είναι μια προσέγγιση που είναι δημοφιλής μεταξύ των ε, επιχειρήσεων. Είναι μια προσέγγιση που ισχύει και σε άλλες απαιτήσεις για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων και των απολογισμών. Η συνένεση που έχει επιτευχθεί για την προσέγγιση συμμορφώσου ή εξήγησε γιατί δεν συμμορφώνεσαι είναι, είναι σωστή και, το είναι μέσα στο πλαίσιο μιας ε, προαιρετικής προσέγγιση. Δεν χρειάζεται λοιπόν να, επιλέξουμε την υποχρεωτική ή την προαιρετική επιβολή αυτών των υποχρεώσεων όπως είχαμε κάνει παλαιότερα όταν ε, ε, η δική μου έκθεση για την εταιρική κοινωνική ευθύνη είχε περάσει στο Κοινοβούλιο είχε συζητηθεί στο Κοινοβούλιο. Τώρα, για το πεδίο εφαρμογή. Πόσο μεγάλη πρέπει να είναι μια εταιρεία ή πόσο πρέπει να είναι ο τζίρο τη ή τι προσωπικό πρέπει να έχει. Ο κύριο Μπαγνιέ έχει υψηλού στόχου. Ε, διπλασίασε τις απαιτήσει σε σχέση με τους υφιστάμενους κανόνες για τις ε, χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η Επιτροπή έκανε και μία αξιολόγηση αντικτύπου. Ε, εμείς από εδώ δεν ξέρω κατά πόσο θα πρέπει να στοχεύσουμε ακόμα υψηλότερα, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλες οι φιλοδοξίες, λίγες είναι οι εταιρείε που θα ενστερνιστούν τα θέματα αυτά. Δηλαδή είναι από τις λίγες φορές που συμφωνώ με την προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πιστεύω ότι και η νομική μας Επιτροπή και η δική μας Επιτροπή θα πρέπει να το υποστηρίξει αυτό. Για το λόγο αυτό, αν καταφέρουμε ε, να το περάσουμε αυτό. Υπάρχουν πάρα πολλές, 36, 49, 78 από τις διάφορες πολιτικές ομάδες θα καταπέσουν. Ε, υπάρχει και μια πρόταση να περάσουμε σε αναφορές στον ετήσιο τζίρο. Εγώ είμαι υπέρ αυτής της προσέγγισης ε, στο πλαίσιο της προσπάθειας επίτευξης συνένεσης. Ο κύριος Ρέτνερ από τους σοσιαλιστές ε, θέλει να εντάξει και κάποια πράγματα για, για τη φορολογία. Εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να πάμε κατά χώρα για τη διαφάνεια στην εκπλήρωση των φορολογικών επιχειρώσεων. Για να είμαι ειλικρινής, επειδή έχω αυτό το φάκελο εδώ και 10 χρόνια, αναρωτιέμαι κατά πόσο είναι χρήσιμο και επικοδομητικό να υιοθετήσουμε αυτή την προσέγγιση κατά χώρα. Εάν η Επιτροπή διαλέξει αυτό το δρόμο θα το στηρίξω. Αναρωτιέμαι όμως μήπως θα έπρεπε να ασχοληθούμε χωριστά με το ζήτημα αυτό και όχι να το συζητήσουμε σε αυτήν την ε, οδηγία η οποία προετοιμάζεται εδώ και τρία χρόνια και έχει ήδη, έχει ήδη συνταχθεί μια μελέτη αξιολόγησης αντικτύπου. Ε, δεν είναι εδώ κανείς ε, για να το συζητήσουμε τώρα. Ε, πολλές από τις τροπολογίες ε, στρέφονται προς την κατεύθυνση της αφαίρεσης του θέματος ε, των απολογισμών σχετικά με φορολογικά θέματα. Η γερμανική κυβέρνηση στην ομάδα εργασίας του Συμβουλίου είναι πάρα πολύ επικριτική για τις προτάσεις αυτές, αλλά ε, είναι διατεθειμένη να ακολουθήσει τον κύριο Μπαρνιέ. Και επίσης και η Business Europe και ο κύριος Μπαλτισάρε στο ΕΛΚΑ έχουν κάνει το ίδιο. Ε, θα ήταν λοιπόν περίεργο εμείς να εμφανιστούμε πιο αρνητικοί απέναντι στην έκθεση από ότι η Business Europe και η γερμανική κυβέρνηση. Θέλω να, να, να πω προς το ΕΛΚ ότι συμφωνώ σε μια συμφωνία ψηφοφορίας μεταξύ ΕΛΚ και Σοσιαλιστών και υποστηρίζω πολλές από τις τροπολογίες τους εκτός από το θέμα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αυτό για μένα είναι ένα ζήτημα αντικρουόμενο. Ε, θα ήθελα να ε, ε, απορριφθούν τροπολογίες οι οποίες προτείνουν τη διαγραφή μεγάλων τμήματων κειμένου όπως και τις τροπολογίες για το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Όπως είπα και την τροπολογία 26 εγκρίνω μεταξύ των τροπολογιών του κ. Μπελόγκ. Νομίζω ότι είχαμε πολύ χρήσιμες ανταλλαγές απόψεων ε, αλλά και ιδίως ε, η προσθήκη του όρου, όπως είπα, where relevant, ε, είναι κάτι που με βρίσκει σύμφωνο. Ελπίζω όμως να κατανοήσουν οι συντάκτες αυτών των τροπολογιών ότι αν συμφωνήσουμε, ο κύριος Ντεβάκ και οι συνάδελφοί του θα πρέπει να αποσύρουν την τροπολογία 20, 36, 37 και 38 76-78 για το πεδίο εφαρμογής και το πρώτο τμήμα της τροπολογίας 79, τροπολογία που η δική μου ομάδα υπέβαλε. Θέλω να σκεφτείτε αν μπορούμε να, στην 43 να διαγράψουμε αυτά για την βιοπικιλότητα και να αποσυρθεί η 58, η 59, η 71, η 84 και η 88 για την προσέγγιση Comply or Explain. Νομίζω ότι οι αποδέκτες της οδηγίας κατανοούν ότι πρέπει να συμμορφωθούν. Δεν είναι ανάγκη να τα κάνουμε πιο αυστηρά τα πράγματα και δεν καταλαβαίνω την, ε, το λόγο της τροπολογίας 67 του κυρίου Ντεμπάκε. Ήδη οι εταιρείε εκδίδουν τέτοιους εκθέσεις και απολογισμούς σε διεθνές επίπεδο και δεν καταλαβαίνω γιατί δεν πρέπει να το κάνουν προς όλους τους συναδέλφους. Έχουμε το θέμα της ε, εφοδιαστικής αλυσίδας, της αλυσίδας αξίας. Ελάχιστοι άνθρωποι αντιμετωπίζουν τα θέματα αυτά με ευθύνη. Και το πρόβλημα δεν αγγείται μόνο σε μια εταιρεία που έχει την καταγεγραμμένη έδρα της σε μια από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τίθενται εδώ και θέματα περιβάλλοντος, επιβολής διακρίσεων κτλ. τα οποία σχεδόν πάντοτε μεταβιβάζονται στην εφοδιαστική αλυσίδα και στην αλυσίδα αξίας. Το να αποκλειστεί λοιπόν η αλυσίδα των προμηθευτών από την ε, οδηγία αυτή ε, δεν πρόκειται να τύχει ευρείας αποδοχής. Από την άλλη γνωρίζουμε ότι υπάρχει μια έντονη ανησυχία ε, αν μια εταιρεία ξαφνικά γίνει υπεύθυνη 100% για κάθε δράση και κάθε προμηθευτή, αυτό θα ήταν απολύτως μη αποδεκτό στις επιχειρήσεις. Υπάρχουν κάποια θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά έχουν βρεθεί απαντήσεις. Πιστεύω ότι οι εταιρείε αξιολογούν και εφαρμόζουν τη δέουσα επιμέλεια, την επιμέλεια που απαιτείται για την επίλυση όλων αυτών των προβλημάτων οι ε, ε, ε, οργανώσεις των εργοδοτών, τα διεθνή επιμελητήρια είναι υπέρ αυτής της προσέγγισης και πιστεύω ότι πρέπει να υιοθετήσουμε κι εμείς μια τέτοια προσέγγιση. Για να είμαι όμως δίκαιος απέναντι στους συναδέλφους Άλντε, οι οποίοι δεν έχουν πιστεί, ε, ως εισηγητής θέλω να τους πω ότι θα δεχθώ τις τροπολογίες τους αν υπάρξει ξεχωριστή ε, ψηφοφορία ως προς τη διατύπωση. Και βέβαια επειδή είμαι ο εισηγητής τους, προφανώς ε, να συνεννοηθούμε και εγώ θα τα συνεννοηθώ όλα μετά με τη γραμματεία. Ίσως θα μπορέσουμε όμως να το συζητήσουμε κι άλλο, γιατί θα ήθελα πάρα πολύ να έχουμε μια συμβιβαστική λύση. Θα το προτιμούσα. Ε, οι συνάδελφοι από το ΕΛΚ είναι πολύ ευτυχείς με την ε, σχετική διατύπωση, οπότε να δούμε και με τον συνάδελφο κύριο Ντεμπάκα. Συγγνώμη που κράτησα το λόγο τόσο πολύ, Πρόεδρε προσπαθώ να καταλήξω σε συμβιβασμούς πάνω σε αυτή την πάρα πολύ σημαντική πρωτοβουλία και θα ήθελα πάρα πολύ να είμαστε θετικοί και επικοδομητικοί για το μέλλον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ αγαπητέ κύριε Ισηγητά. Δυστυχώς ε, ε, απουσιάζουν οι περισσότεροι στους οποίους αναφερθήκατε. Ελπίζω πάντως οι παρόντες να βοηθήσουν ε, τους απόντες να συμφωνήσουν μαζί σας, τουλάχιστον να να συμπλέψουν κάποια στιγμή. Ζήτησαν το λόγο ο κύριος Ντεπάκερ και μετά η Τζέιν Λάμπερτ. Ο Φίλιπ Ντεπάκερ πρώτα και μετά ο κύριος Ρέινερ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τον συγητή για τις εργασίες του και τις εκτεταμένες εξηγήσεις που μας έδωσε και βεβαίως για την ε, επικοδομητική συζήτηση που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο. Νομίζω ότι κατακτήσαμε κάποια πρόοδο, κάναμε κάποιους συμβιβασμούς ε, για τα ζητήματα που, στα οποία αναφέρθηκε και στην εισαγωγή του. Συνειδητώ επίσης ότι είναι πολύ σύνθετα και κάπως συναισθηματικά τα ζητήματα αυτά. Ε, πολλές τροπολογίες προτάθηκαν και είναι δύσκολο βεβαίως ε, να καταλήξουμε σε συμβιβασμό όταν ε, κοιτάξει κανείς όλες τις τροπολογίες από τα αριστερά, από τα δεξιά και να διασφαλίσει κανείς ότι θα πρέπει να είναι αποδεκτές από όλους. Να ξεκινήσω με το συμμορφώ σου ή σου. Νομίζω ότι έχει δίκιο ο εισηγητής. Αν ζητούμε από τις εταιρείες είτε να συμμορφώνονται είτε να ε, δώσουν εξηγήσεις, τότε θα πρέπει να δίνουν λόγω γιατί δεν ε, συμμορφώνονται. Μπορούμε λοιπόν να κάνουμε κάποια πρόοδο. Θα ξαναπροσπαθήσουμε με την ομάδα μου να επανέλθουμε για να βρούμε έναν καλό συμβιβασμό και να βρούμε μια καλή διατύπωση. Κάποιοι από τους συναδέλφους μας επίσης ε, πρότειναν τροπολογίες για το πεδίο. Ε, είναι υπέρ ενός λιγότερο ευρέως πεδίου. Ο εισηγητής αντίθετα ε, θέλει ένα ευρύτερο πεδίο. Νομίζω ότι το σημαντικότερο είναι να ορίσουμε στο πεδίο ποιες εταιρείε εμπίπτουν στον κανονισμό. Θα συμπεριλαμβάνονται βεβαίως και οι μεγάλες εταιρείες, αλλά αν πρέπει να ε, πάμε και στις μικρότερες, τότε θα πρέπει και νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε έναν συμβιβασμό. Και δύο ακόμη σημεία που θα ήθελα να πω. Ένα για τον ε, συμβιβασμό C έχετε ε, την, ε, την αναλογία ανάπηρων ατόμων και τα λοιπά. Νομίζω ότι δεν είναι πολύ ρεαλιστική αυτή η προσέγγιση. Βεβαίως μια εταιρεία μπορεί να έχει μια γενική προσέγγιση για το πώς ε, αντιμετωπίζει ε, ανθρώπους με αναπηρίες, ε, ανθρώπους με, που προέρχονται από μειονότητες. Ταυτόχρονα όμως δεν μπορούν οι εταιρείε όταν του προσλαμβάνουν να του ζητούν πληροφορίε για αναπηρίε ή για το υπόβαθρό του, για την προέλευσή του. Από αυτή την άποψη νομίζω ότι θα πρέπει να αλλάξουμε κάπω τη διατύπωση, ώστε βεβαίω να ζητούμε από τι εταιρείε να έχουν μια ευρύτερη αντίληψη, αλλά λαμβάνοντα υπόψη ότι υπάρχει και μια πυκλομορφία όσον αφορά τις, ε, τα δικαιώματα του τι μπορούν να ζητούν, να ρωτούν τους ανθρώπους. Τέλος, Πολύ σημαντικό σημείο για μας. Για να μην πω κρίσιμο, αφορά την, την ε, αλυσίδα αξίας. Είχαμε αυτή τη συζήτηση στη συνάντηση των σκιωδών ε, εισηγητών είχαμε πει ότι είναι πολύ δύσκολο να το αποδεχτούμε διότι ως έχει μιλούμε για ολόκληρη την αλυσίδα άξιας και νομίζω ότι δεν είναι αυτή η λύση που θέλουμε να, στην οποία θέλουμε να καταλήξουμε. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Αν δείτε το μολύβι, ένα μολύβι ε, έχουν συνήθως αυτή τη σβίστρα. Θα διασφαλίσουμε δηλαδή ότι η εταιρεία που φτιάχνει το μολύβι θα πρέπει να ελέγχει όλη την αλυσίδα της, ακόμα και αυτόν που φτιάχνει την σβιστρούλα. Νομίζω ότι είναι υπερβολικά μεγάλο το, το άχθος για τις εταιρείε. Είναι πολύ, πολύ, νομίζω, δεν, αμφιβάλλω αν αυτή είναι η καλύτερη λύση. Είναι πολύ δύσκολο το σημείο αυτό. Συζητήσαμε βεβαίως και την προηγούμενη εβδομάδα στη συνάντηση των σκιωδών νησιωτών. Προσπάθησα να τους ε, να πείσω του συναδέλφου, μου, αλλά για μας εξακολουθεί να είναι ένα πολύ δύσκολο ζήτημα αυτό, οπότε ενδεχομένω και ο εισηγητή μπορεί να κάνει κάτι προς αυτή την κατεύθυνση. Πάντω, αν πάει έτσι την ψηφοφορία, για μας θα είναι πολύ δύσκολο να το υποστηρίξουμε. Και ζητώ και από τους συναδέλφου, ε, τους υπόλοιπους συνελεύους να ε, το λάβουν υπόψη σε αυτό. Λοιπόν, να συνοψίσω. Βεβαίως έχουμε κάνει πρόοδο, έχουμε αποκλίνουσες απόψεις για το φάκελο αυτό. Κάποια ζητήματα εκκρεμούν ακόμη, όπως είπε και ο εισηγητής, αλλά νομίζω ότι μέχρι στιγμής έχουμε συνεργαστεί με ανοιχτό πνεύμα και ελπίζω το ίδιο να ισχύσει και τις επόμενες μέρες και εβδομάδες και να καταλήξουμε σε μια συμφωνία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Ντεμπάκερ. Φαίνεται ότι όλοι αρχίζουμε να αποκτούμε κακές συνήθειες όλοι αρχίζουμε και παραβαίνουμε το χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας. Εντάξει, είμαστε επικείς με το συντάκτης γνωμοδότης, αλλά οι υπόλοιποι ομιλητές θα πρέπει να είναι πιο συνέπει ε, στην ε, τήρηση του χρόνου. Δεν θέλω να σας λογοκρίνω, αλλά λίγη προσοχή. Κυρία Ρέινερ, ε, τι γίνεται με τον Τζαμπαόρη. Απουσιάζει η κυρία Ράινερ και μετά η κυρία Σαϊά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω δεν θα με μαλώσετε εμένα, θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Ο Ρίτσαρτ Χάουιτ είπε πάρα πολλά πράγματα, τα οποία θέλω κι εγώ να υποστηρίξω. Να πω όμως τα εξής. Η έκθεση αυτή είναι πολύ σημαντική από πρακτικής άποψης για την πρακτική οικονομική ζωή. Μίλησα και με πολλού εκπροσώπους επιχειρήσεων και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό η Επιτροπή μα να ε, ε, λάβει μια πολύ συγκεκριμένη ε, θέση για τις τροπολογίες. Για μένα ήταν πολύ σημαντικό ο, να μειωθεί ο αριθμός των υπαλλήλων που είναι απαραίτητος για την υποβολή έκθεσης. Και αυτό διότι με απελπισία βλέπω πως στην, του, Ολομέλεια του Κοινοβουλίου συζητήσαμε για τα εργοστάσια που κάηκαν στον, Παγκλα... στο όπου έχουμε εταιρείε οι οποίες δεν αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους και ο Ρίτσαρτ Χάουιτ όχι μόνο σε αυτή τη θητεία αλλά και στο παρελθόν ε, ήταν πολύ αξιόπιστος ως προς τις ε, ε, εισηγήσεις του και μας έδειξε ότι πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας όχι μόνο όταν οι εταιρείε είναι πολύ μεγάλες Είμαι πρόθυμη λοιπόν να καταλήξουμε και σε συμβασμούς όσον αφορά τις τροπολογίες μου. Αλλά για παράδειγμα είπα ότι χρειαζόμαστε περισσότερο ε, φως ε, και ως προς τις, τους μισθούς και πόσο υπεύθυνε ή ανεύθυνες είναι οι εταιρείε. Αυτά ήθελα να πω για τις ε, τροπολογίες μου όσον αφορά τα φορολογικά θύματα οι συμβιβασμοί είναι καλοί, αλλά και ολόκληρο το πακέτο μέτρων θα πρέπει να είναι σωστό και κατάλληλο. Η ε, κυρία Εσάια. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή μας τον κύριο Χόουιτ για την πολύ καλή δουλειά του και να επισημάνω ορισμένα ζητήματα. Γιατί το ΕΛΚ και ως ομάδα αλλά και πολλοί μεμονωμένοι βουλευτές δεν είναι κατά της ε, αρχής της διαφάνειας Αλίμονο, συμφωνούμε πλήρως με την αρχή της διαφάνειας. Επίσης, ε, η ενημέρωση για μη χρηματοοικονομικά θέματα είναι καλό και για τις ε, επιχειρήσεις. Να πούνε ότι αυτή είναι η πηγή των ε, προϊόντων μας, έτσι γίνονται. Αυτό είναι πολύ, αυτός ο απολογισμός είναι πολύ θετικός και για τις εταιρείε. Όταν όμως επιμένουμε σε μη χρηματοοικονομικές πληροφορίες, θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι θα, μπορούμε, θα μπορεί να γίνει εξακρίβωση. Αν ζητούμε στον ετήσιο απολογισμό να λένε οι εταιρείε πώς ε, σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, εντάξει να πούμε κατά πολέμηση διαφθοράς, αλλά το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή θέματα συναφή με τους ε, εργαζόμενους, όπως είπε ο συνάδελφος από του φιλελεύθερου, πώς ε, οι ελεγκτές θα εξακριβώσουν την αλήθεια αυτή της ετήσια έκθεσης, Κάποιο θα κρίνει ότι όντω αυτή η εταιρεία σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα στην παραγωγή της. Ποιο είναι το κριτήριο αυτού του ελέγχου, αυτής της εξακρίβωσης, γιατί σε πολλές χώρες έχουμε τέτοια νομοθεσία ε, ε, ελέγχου, αλλά όταν περιλαμβάνουμε κάποιο στοιχείο στον ετήσιο απολογισμό θα πρέπει να επιδέχεται εξακρίβωσης. Τώρα να λέμε όπου είναι δυνατό να αποκλείεται από τον έλεγχο. Γιατί μπορούμε να ζητήσουμε να γίνεται έλεγχος για ορισμένα πράγματα που όμως δεν είναι ελέγξιμα εκφύσεως. Οπότε και οι επιθεωρητές, οι ελεγκτικές εταιρείες πολύ απρόθυμα θα κάνουν δηλώσεις για πράγματα που δεν μπορούν να εξακριβώσουν αν όντως ισχύουν. Μπορούν απλώς να λένε ότι ελπίζουμε ότι η εταιρεία αυτή πληρεί τις προϋποθέσεις ε, που ισχυρίζεται, ότι σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα για παράδειγμα, αλλά από τη στιγμή που δεν μπορούμε να το εξακριβώσουμε αυτό, είναι κάπως περίεργη κατάσταση, παράδοξη. Και κάτι άλλο, συναφές με το προηγούμενο. Όταν λέμε να γίνεται περιγραφή των ε, βασικών κινδύνων, στον έλεγχο δεν υπάρχει περιθώριο για ε, προβλέψεις για μαντίες. Θα πρέπει να υπάρχει βεβαιότητα, όχι απλώς εικασίες. Αν ο ελεκτής δεν είναι βέβαιος, δεν λέει τίποτα. Τώρα, μόνο ουσιαστικές πληροφορίες που μπορούν να ελέγχονται, να περιλαμβάνονται στον ετήσια έκθεση, στον ετήσιο απολογισμό. Να βρούμε τη σωστή διατύπωση για να ξεπεράσουμε αυτό το πρόβλημα. Γιατί στις σκανδιναβικές χώρες έχουμε πολύ αυστηρές νομοθεσίες για τον έλεγχο και θα πρέπει να ελέγχονται τα ζητήματα που περιλαμβάνονται στο, στην ετήσια έκθεση. Και κάτι άλλο, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είπατε ότι αυτά τα στοιχεία προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ότι υπάρχει μελέτη που θεμελιώνει αυτά τα στοιχεία. 500 εργαζόμενοι όμως είναι μεγάλος αριθμός. Και όταν έχουμε 20 εκατομμύρια ευρώ στο συνολικό ισολογισμό και 40 εκατομμύρια ετήσιο τζίρο, αυτό δεν είναι και πολύ μεγάλο το νούμερο. Οπότε διαρωτώ με μήπως έτσι προσθέσουμε άχθος γραφειοκρατικό στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αν μπορούμε να βρούμε κάποια συμβαστική λύση, αν ελαφρύνουμε να απαλλάξουμε κάπως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Άλλωστε, είπατε ότι θα φροντίσετε να αποφευθεί το περαιτέρω άχθος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γιατί είμαι βεβαίω ότι και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θέλουν να, να για τα θετικά στοιχεία της αλυσίδας παραγωγής τους. Οπότε μπορούμε να είμαστε βέβαιοι για την καλή τους θέληση πολύ ευχαρίστω θα δηλώσουν τέτοια πράγματα. Αυτά και ελπίζω να ληφθούν υπόψη και οι δικέ μα ανησυχίε. Σα ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελε το λόγο. Παρακαλώ. Ε, χρόνου φίδου, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Όντω είμαι λακωνικό. Θα ήθελα να σα υπενθυμίσω ότι εκτιμώ ιδιαίτερω τι προσπάθειε τη Επιτροπή σα και χαίρομαι για την πρόοδο που έχετε σημειώσει μέχρι τώρα, που άλλωστε οδεύει προς τη σωστή κατεύθυνση. Άλλωστε δεν ήταν περίεργο που στην αρχή είχαμε διάσταση απόψεων. Πάντως ε, φαίνεται ότι πάμε προς το σωστό δρόμο πια. Κάποια τεχνικά σχόλια που ίσως βοηθήσουν. Καταρχήν για το πεδίο εφαρμογή. Πρόθεση μας ήταν να βρούμε μια ισορροπία και εντοπίσαμε τον αριθμό των εργαζομένων ως βασική παράμετρο για να ε, κρίνουμε τη σημασία της ε, σχετικής ενημέρωσης. Επίσης αναφέρθηκαν ε, ανησυχίες για, τις, για τα στοιχεία του ισολογισμού ή του ετήσιου τζίρου, αν είναι αρκετά υψηλά. Πάντως η υποχρέωση δημοσιοποίησης έχει τέτοια δομή ότι αν ώστε μία οτι αν μια επιχειρηση που δεν θα έχει 500 εργαζομένους δεν θα υπόκειται στην υποχρέωση τέτοιες παροχής πληροφορίας γιατί πρώτα θα πρέπει να εκπληρωθεί το, το κριτήριο του αριθμού των εργαζομένων και μετά του τζίρου και του ισολογισμού. Αν δεν ε, εκπληρωθεί το πρώτο κριτήριο των εργαζομένων δεν υπάρχει καν υποχρέωση, δεν υπάρχει η εταιρεία υποχρέωση ε, παροχής ε, του, ισολο, του απολογισμού. Επίσης, 18.000 εταιρείες είναι περίπου ο στόχος της πρότασης και με το κατόφλι των 250 εργαζομένων θα είχαμε αύξηση του αριθμού των εταιριών σε 42.000 από 18. Και μέχρι στιγμής 2.500 εταιρείες κάνουν τέτοια ενημέρωση. Πάντως χαίρομαι που ασχοληθήκατε και με το θέμα της αλυσίδας ενεφοδιασμού. Είναι πολύ σημαντικό θέμα. Δεν ε, εμπίπτει βέβαια στην πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής εμέσως ε, γινόταν αναφορά αυτού του θέματος μέσω των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της διαφθοράς και της προστασίας του περιβάλλοντος. Πάντως άμεσα δεν υπήρχε τίποτα για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. ο κύριος συγγετής και πάλι. Ελπίζω ότι οι εξηγήσει ε, ε, βοηθούν να κατευναστούν οι ανησυχίες των άλλων μελών. Ε, θα υπάρχουν πάρα πολλοί... Ε, ε, εγώ θα υποστηρίξω όλες τις τροπολογίες που κάνουν, καθιστούν σαφές το κείμενο. Για το θέμα της ποικιλομορφία. Συμφωνώ απολύτως. Το θεωρώ ως ένα ζήτημα στο οποίο, γύρω από το οποίο μπορεί να βρεθεί συμβιβασμός. Ε, κατά εμέ είναι απολύτως δυνατόν για τις επιχειρήσεις να έχουν ε, ε, πολιτικές προσλήψεων που θα θέτει τα ίδια κριτήρια και ότι θα εντάσσουν όλες τις κοινωνικές ομάδες. Πάνω στο θέμα αυτό είμαι σίγουρος ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε συμφωνία και σε συμβιβασμό για την αλυσίδα αξία, την, αλυσίδα των προμηθευτών. Σε ευχαριστώ για αυτό που είπες και, και, τις δύο σας ευχαριστώ, ιδίως την κυρία Χάιερ. Πράγματι υπάρχει ένα μεγάλο ακροατήριο επιχειρήσεων που παρακολουθούν αυτή τη συζήτηση και είναι σημαντικό να στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα και να πούμε ότι επί της αρχής συμφωνούμε. Έχω συζητήσει ε, με τον κύριο Ντεμπάκερ, έχει και εκείνος ε, κουβεντιάσει με τις επιχειρήσεις θα είναι πιο εύκολο για μας ε, εδώ στο Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή μας ε, να μας μεταφερθούν τα σχόλια αυτά από τον επιχειρηματικό κόσμο. Ε, βέβαια σέβομαι την προσέγγιση της Άλντε. Ε, εν τέλει θα ζητήσω ξεχωριστή ψηφοφορία όπως είπα. Οπότε οι απόψεις της Άλτε θα περάσουν. Ε, βεβαίως το πεδίο εφαρμογής θα μπορούσε να διευρυνθεί και να συμμετέχει μεγαλύτερος αριθμός επιχειρήσεων. Ε, εσείς αναφερθήκατε ε, στα συστήματα ελέγχων. Ε, προσπαθώ να επιτύχω μια, ένα συμβιβασμό εδώ πέρα και για τις δύο πλευρές. Στην κυρία Χέιεν ε, ε, για, τη, για τις χώρες Έχετε κάνει μια τροπολογία για, για ένα διπλό σύστημα δημοσίευσης εκθέσεων και αναφορών. Οι επιχειρήσεις δεν το επιθυμούν αυτό. Ε, παρακαλώ να το σκεφτείτε. Ε, δεν πρόκειται να υπάρξει ένας έλεγχος επί αυτών των εκθέσεων και των αναφορών όπως είναι ο οικονομικός έλεγχος. Ε, οι ελεγκτικές αρχές έχουν ε, ε, εξειδικευμένα τμήματα τα οποία ελέγχουν και αναφορές σχετικά με την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Νομίζω ότι δεν είναι αδύνατον. Πιστεύω ότι ο κύριος Μπαρνιέ έχει βρει μια πολύ επιτυχημένη ε, συμβιβαστική λύση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποστήριξή σας. Ευχαριστούμε κύριε Σιγητά. Να σας υπενθυμίσω ότι οι συμβαστικές τροπολογίες ε, θα ψηφιστούν πρώτα ε, οι προτάσεις διαγραφής και μετά οι υπόλοιπε. Δεν θα συμβεί αυτό που έγινε στην προηγούμενη ψηφοφορία. Και επίσης ε, δεν έχουμε ψηφοφορίες κατά τμήματα σε μια συμβαστική λύση. Μια συμβαστική λύση είναι συμπαγή, την ψηφίζουμε ακέραιη, όχι κατά τμήματα. Αύριο θα ε, ψηφίσουμε εμείς, ώστε η Νομική Επιτροπή να συμπεριλάβει τις προτάσεις μας την ψηφοφορία της βασικής έκθεσης που θα γίνει 17 Δεκεμβρίου. Ωραία, ολοκληρώσαμε αυτό το θέμα και περνάμε στο σημείο 4, στην έκθεση Steinruck. Θα μας παρουσιάσει τις συμβαστικές τροπολογίες ε, επί της εκθέσεως πρωτοβουλίας για τις πραγματικές επιθεωρήσεις εργασίας ως στρατηγική για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στην Ευρώπη. Κυρία Στάιμπρουκ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πριν από λίγα λεπτά ήμουν ακόμη πεισμένη ότι θα καταφέρναμε να υποβάλουμε μια καλή εισήγηση προς όφελος των νόμιμων εταιρετών, των εταιριών και των υπαλλήλων που ε, πλήττονται από την ε, κατάχρηση, από την παραβίαση μάλλον της νομιμότητας. Είχαμε συνάντηση σκιωδών, εισηγητών και συζητήσαμε πολύ έντονα για συμβαστικές προτάσεις. Έκανα κινήσεις υποχώρησης προς όλες τις πολιτικές ομάδες. Δεν έγιναν αποδεκτές οι προσπάθειες μου από και θέλω να τονίσω ξανά. Δεν θέλω να υπησέλθω ούτε σε αρμοδιότητες των κρατών μελών, ούτε να βλάψω ε, επιχειρήσεις. Σκοπός μου είναι ακριβώς να ενισχύσουμε τις επιχειρήσεις και τα κράτη-μέλη και η έκκλησή μου είναι σήμερα στη συζήτησή μας να μην χάσουμε καμία ευκαιρία για ζητήματα όπου θα μπορούμε πραγματικά να καταλήξουμε σε κοινή θέση της ε, Επιτροπής με συγκεκριμένο και σαφές μήνυμα ότι δεν θέλουμε παρανομία και κατάχρηση στην Ευρώπη. Και νομίζω ότι θα έπρεπε να είμαστε στη θέση να φτάσουμε ε, σε συμβιβασμούς. Η εισήγηση είναι απαραίτητη αφού γνωρίζουμε ότι η μαύρη εργασία αυξάνεται στην Ευρώπη τρομακτικά ε, φοροδιαφυγή και κατάχρηση εργαζομένων. Οι επιθεωρήσεις εργασίας μειώνονται τρομακτικά. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι εργάζονται σε επισφαλείς σχέσεις εργασίας. Ιδιαίτερα όταν είναι μετακινούμενοι εργαζόμενοι. Ιδιαίτερα σε ε, αλυσίδες υπεργολαβίες και γι' αυτόν τον λόγο μόνο ευρωπαϊκά μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα αυτό. Μίλησα με κράτη-μέλη, πολλά. Και είμαι πεπισμένη. Είναι πολύ δύσκολο να παρακολουθήσουν 7 και 8 υπεργολάβους. Και στην Επιτροπή μας είχαμε συζητήσει και νωρίτερα, ε, παλαιότερα, για μια υπόθεση στο Φλαμανβίλ. Κλασικό παράδειγμα περίπτωσης όπου θα ε, ήταν αναγκαίες κοινέ επιχειρήσεις, κοινή έλεγχη για εταιρείε ε, ταχυδρομικές θερίδες κτλ. Υπάρχουν από μεγάλη πολιτική ομάδα μεγάλες επιφυλάξεις όσον αφορά την συμπερίληψη των κοινωνικών εταίρων. Να θυμίσω και σε αυτό το ζήτημα. Υπάρχουν κράτη-μέλη όπου αυτό είναι το ισχύον δίκαιο. Και το είχαμε συζητήσει και εδώ, ότι και οι κοινωνικοί εταίροι ε, και τα συνδικάτα ενδιαφέρονται για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας και για την τήρηση των νόμων. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο υπάρχουν τόσο μεγάλα προβλήματα με αυτή την εισήγηση ακριβώς επειδή στο ένα ή στο άλλο μέρος της ε, αναφέρονται και οι κοινωνικοί εταίροι, δηλαδή η πραγματικότητα που ισχύει σε πολλά κράτη-μέλη. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να ενισχύσουμε ε, αυτή την εισήγηση, ε, νόμιζα δηλαδή ότι θα μπορούσαμε, αλλά από ό,τι βλέπω θα πρέπει να συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις μέχρι αύριο και θα δούμε αν είναι κενό γράμμα το να υποστηρίξουμε τα φορολογικά έσοδα των κρατών μελών και όχι μόνο να ζητούμε νέους φόρους και αν πράγματι ενδιαφερόμαστε για την προστασία των εργαζομένων όταν υπάρχουν διαμεσολαβητές οι οποίοι εκμεταλλεύονται παράνομα ανθρώπους. Το μόνο που θέλουμε να επιτύχουμε είναι η κατάργηση της ε, παράνομης εκμετάλλευσης και γι' αυτό το λόγο ως Κοινοβούλιο είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μια ολοκληρωμένη και καλή θέση για το ζήτημα αυτό. Μάλιστα. Δεν βλέπω κανένα ζητάει το λόγο. Α, ο κύριος ε, Όρη. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Δυστυχώς η μα η βρίσκεται σε μια κοινοβουλευτική αποστολή εκτό ε, Βρυξελών. Δεν θα ήθελα εδώ να τον αναπληρώσω, αλλά να μιλήσω ω ε, τσαμπαόρι. Θα δώσω την προσωπική μου γνώμη. Έχω κάποια προβλήματα με την τελευταία εκδοχή των συμβαστικών τροπολογιών. Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Για τη συμβαστική τροπολογία σιγματάφ, F. Το πρώτο πρόβλημα που έχω είναι με την ε, συμβαστική τροπολογία F. Γιατί ε, έχω πρόβλημα με την παράγραφο που μιλάει για τα συλλογικά δικαιώματα. Πρόκειται για μία Συζήτηση που γίνεται σε πολλές χώρες εδώ και πολύ καιρό. Με διαφορετικές πρακτικές και παραδόσεις. Και για τις ε, ενώσεις εργαζομένων, εργοδοτών και για τα συνδικάτα. Μερικές φορές τα συνδικάτα δεν εκπροσωπούν όλους τους εργαζόμενους. εξαρτάται από το εύρος της εντολής τους. Οπότε θα πρέπει να αλλάξουμε κάπως την διατύπωση της συμβαστικής τροπολογίας ΣΥΓΜΑΤΑΒ, γιατί τα συστήματα, επαναλαμβάνω, διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Γι' αυτό και θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Δεύτερο θέμα, συμβαστική τροπολογία J που μιλάει για εκ των υστέρων εγγραφή. Πώς θα γίνει αυτό στην πράξη. Εκ των υστέρων καταγραφή. Ποιες είναι οι πληροφορίες που θα πρέπει εκ των προτέρων ή εκ των υστέρων να χορηγεί ο εργοδότης στην επιθεώρηση εργασίας. Συμβαστική τροπολογία ε. Αυτή και αν είναι προβληματική. Εκεί λέμε ότι οι εκπρόσωποι των εργαζομένων παρεμβαίνουν σε μια επιθεώρηση εργασίας. Διαφωνώ ριζικά. Θεωρώ ότι η επιθεώρηση εργασίας θα πρέπει να γίνεται αυτόνομα από τις αρχές. Οι αρχές στην περίπτωση αυτή είναι υπεράνω και των εργαζομένων και των εργοδοτών φυσικά υπόκεινται στον νόμο αυτές οι επιθεωρήσεις εργασίας. Το να συμμετέχουν τώρα στις ε, φορείς επιθεωρήσεις εργασίας, είτε εργαζόμενοι είτε εργοδότες, είναι απαράδεκτο και δημιουργεί σοβαρά προβλήματα και διαχείρισης. Δεν μπορεί ταυτόχρονα να κανείς να είναι και δικαστής και κατηγορούμενος. Δεν είναι δυνατόν να περιμένουμε αντικειμενικότητα από ανθρώπους που κρίνουν αυτούς σε τελική ανάλυση. Και αυτό θα συμβεί αν εκπρόσωποι των εργοδοτών ή των εργαζομένων συμμετέχουν στις επιθεωρήσεις εργασίας. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον κατώτατο μισθό ή και το ίση αμοιβή για ίση εργασία. Είναι θέματα αρχής εδώ. Μπορεί να συμφωνούμε ή να διαφωνούμε, δεν θα επαναλάβουμε την όλη συζήτηση είπαμε ότι αυτό θα, το κρίνουν οι αγορές. Αλλά τώρα να είναι η μισθή αντικείμενο εξέταση από την επιθεώρηση εργασίας, αυτό είναι απαράδεκτο. Οι επιθεωρήσεις εργασίας θα κρίνουν αν ε, τηρούνται οι νομοθετικές διατάξεις από τις επιχειρήσεις. Οι διατάξεις του εργατικού δικαίου. Τώρα, να συμπεριλάβουμε στο πεδίο ελέγχου των επιθεωρήσεων εργασίας και την ε, εξέταση συγκεκριμένων συμβολέων και όρων συμβολέων όπως είναι η μισθή είναι απαράδεκτο. Επίσης και το συμβαστική τροπολογία ΚΑΠΑ αφήνει τεράστιο πεδίο στις επιθεωρείς εργασίες και ουσιαστικά τις φέρνει στην ε, ιδιωτική σφαίρα των ε, εργοδοτών. Νομίζω ότι είμαστε υπερβολικοί στο σημείο αυτό. Θεωρώ ότι μπορούμε να βρούμε μια πιο λογική λύση. Τώρα, συμβαστική τροπολογία λάμδα. Το μείζον πρόβλημα που έχουμε την τροπολογία αυτή αφορά για ανθρώπους που έχουν κάνει ψευδείς δηλώσεις. Θα θυμάστε τις φοδρές συζητήσεις είχαν γίνει στην αρχή της κοινοβουλευτικής θητείας για το θέμα αυτό ιδιαίτερα όταν μιλούσαμε για το ωράριο εργασίας των ε, φορτηγατζίδων. Τώρα, όταν έχουμε έναν εργαζόμενο από κοινωνικής απόψεως, που στην ουσία είναι αυτοαπασχολούμενος ή ψεύτο ανεξάρτητος, και αυτό το θέμα ορισμού του ψευδοανεξάρτητου επιχειρηματία είναι δύσκολο. Τώρα να περιμένουμε ότι οι επιθεωρείς εργασίας ε, θα διαλευκάνουν θέματα για τα οποία εμείς δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε για τον ορισμό τους είναι υπερβολικό. Συμβαστική τροπολογία μη. Εκεί αναφέρονται οι αρχές εργασίας. Οι αρμόδιοι φορείς. Εδώ μιλούμε για εθνικές αρμοδιότητες. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις διατάξεις ε, περί μετανάστευσης, αυτά τα θέματα είναι εθνικά, εθνικής αρμοδιότητας. Δεν μπορούμε να περιμένουμε από την ε, επιθεώρηση εργασίας ε, να κάνει παρατηρήσεις σχετικά με τους όρους υποδοχής των μεταναστών από ένα κράτος μέλος. και η συμβαστική τροπολογία μου δημιουργεί πρόβλημα. Και υπάρχει εδώ ένα γενικότερο πρόβλημα. Το αναφέραμε και προηγουμένως, όταν αναφερθήκαμε στην οδηγία για τους αποσπασμένους εργαζόμενους. Μερικές φορές, ακόμη και με ένα κόμμα ή μία τελεία, φαίνεται να βάζουμε στο ίδιο τσουβάλι τους διακινητές και τους ελαφρομετανάστες. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να εξομοιώνουμε τις κατηγορίες αυτές. Συμβαστική τροπολογία όμικρον. Και με αυτήν έχω πρόβλημα. Τι κατάρτιση προτείνεται εδώ. Μιλούμε για τους αποσπασμένους εργαζόμενους, ε, τους ε, μετανάστες. Αυτά τα ζητήματα δεν είναι κοινοτική αρμοδιότητα, αλλά εθνική. Κάθε χώρα θα αποφασίσει τι κατάρτιση χρειάζεται για να διορθωθούν τα προβλήματα που έχει. Συμβαστική τροπολογία Z, τελευταία. Το ίδιο και εδώ ισχύει. Έχουμε εθνικές αρμοδιότητες. Δεν μπορούμε λοιπόν να έχουμε ελάχιστους ευρωπαϊκούς κανόνες για την επιθεώρηση εργασίας, γιατί το θέμα αυτό δεν εμπίπτει στις κοινοτικές αρμοδιότητες, αλλά είναι εθνική αρμοδιότητα. Συμβαστική τροπολογία ΕΕ. Μερικές φορές έχω την αίσθηση ότι φτάνω μέχρι τα όρια της ξενοφοβίας όταν μιλούμε συστηματικά για κοινωνικό ντάμπινγκ. Σαν να θεωρούμε οποιοδήποτε τρίτο που έρχεται στη χώρα μας ότι θα ασκήσει κοινωνικό ντάμπικ στη χώρα υποδοχής. Αυτή η ισορροπία έχει μερικές φορές επιζήμιες συνέπειες, απαράδεκτες. Πιστεύω ότι θα πρέπει να αναζητήσουμε λύσεις για να σημειώσουμε πρόοδο και να σεβαστούμε τις εθνικές αρμοδιότητες Πιστεύω ότι μπορούμε να βρούμε λύσεις. Για παράδειγμα, βέλτιστες πρακτικές, ανταλλαγή καλών πρακτικών, η των πρακτικών μεταξύ των χωρών μελών. Έτσι θα κάνουμε αναλύσεις ε, των καλών πρακτικών των άλλων χωρών και θα αντιλήσουμε κάποια συμπεράσματα. Ο ορισμός των προβλημάτων, η σωστή διάγνωση είναι πολύ σημαντικά θέματα. Αλλά τώρα να έχουμε προσδοκίες ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο χωρίς να υπάρχει κοινοτική αρμοδιότητα είναι υπερβολικό. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να συμπληρώσω δύο θέματα εδώ. Μερικές ομάδες πολιτικές είναι κατά της ιδέας της, της κάρτας κοινωνικής ασφάλισης των διακινούμενων εργαζομένων. Κάτι που θα διευκόλυνε το έργο των επιθεωρητών εργασίας. Πώς είναι δυνατόν να διαφωνεί κανείς με μια τέτοια ευρωπαϊκή ασφάλιση. Άλλωστε, ήδη στην οδηγία για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων υπήρχε κάτι αντίστοιχο. Και αυτή η ιδέα της Ευρωπαϊκής Κάρτας Κοινωνικής Ασφάλισης ήταν και μάλιστα πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κατάλαβα ότι ακόμη και οι πράσινοι έχουν πρόβλημα, αλλά δεν αντιλαμβάνομαι γιατί. Γιατί αν η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς συμφώνησε μεγάλη πλειοψηφία για τη θέσπιση αυτής της Ευρωπαϊκής Κάρτας Κοινωνικής Ασφάλισης και μάλιστα είχαμε και τη συμφωνία του Συμβουλίου, γιατί είναι ουσιαστικά μια κάρτα που διευκολύνει την επαγγελματική κινητικότητα. Και αυτό το κάναμε για τα επαγγελματικά προσόντα. Γιατί να μην έχουμε μια αντίστοιχη κάρτα κοινωνική ασφάλιση και εμεί. Δεν καταλαβαίνω τα... τις ομάδες που είναι κατά. Επίσης έτσι θα μπορούσαμε να έχουμε μια, έναν ευρωπαϊκό φορέα, μια ευρωπαϊκή ελίτ που θα ε, εγκύπτει οριζόντια σε κάποια προβλήματα που αφορούν τις εργασιακές συνθήκες ε, ανεξάρτητα για ποιον τομέα μιλάμε. Και αυτό δεν εμποδίζει σε καμία περίπτωση την επικουρικότητα, ούτε σφετερίζεται εθνικέ αρμοδιότητε. Εν πάση περιπτώσει, κύριε Σιγήτρη, έχετε το λόγο. Ναι. Νομίζω ότι η συζήτηση γίνεται σε πολύ ιδεολογική βάση και δεν λαμβάνει υπόψη τις πραγματικότητες που έχουμε στην ε, Ευρώπη η εργασιακή μετανάστευση, η απόσπαση εργαζομένων, η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων σε όλα τα κράτη-μέλη, να εργάζονται σε όλα τα κράτη-μέλη. Είναι δεδομένη, είναι διασφαλισμένη, αλλά γνωρίζουμε ότι υπάρχουν, δημιουργεί και κάποια προβλήματα όπου υπάρχουν νομικά κενά και στα κράτη-μέλη ή εκεί όπου υπάρχει ανεπαρκές προσωπικό, υπάρχουν και διαφορές ε, των διοικητικών δομών που επίσης δημιουργούν ορισμένα προβλήματα. Πραγματικότητα είναι, και το είπα και στην αρχή της συζήτησής μου, ότι έχουμε πολλά δισεκατομμύρια χρημάτων που χάνονται από τη φορολογία στα κράτη-μέλη. Ιδιαίτερα στα κράτη-μέλη που διέρχονται οικονομικά προβλήματα τα οποία θα μπορούσαν αντί να αυξάνουν τους φόρους για τους υπαλλήλους και τις επιχειρήσεις να καταπολεμήσουν την ε, παρανομία. Και βεβαίως δεν είναι παράνομος όποιος ε, ε, μεταβαίνει σε διαφορετικές χώρες το συμφωνούμε σε αυτό, αλλά έχουμε πάρα πολλά προβλήματα ακόμη και εμπορία ανθρώπων στην Ευρώπη που αποδεικνύουν ότι πρέπει να καταπολεμηθούν οι παραβιάσεις. Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε προβλήματα σε επιχειρήσεις που είναι νόμιμες ή ακολουθούν την, ε, τους νόμους. Το αντίθετο, να καταπολεμήσουμε τις παρανομίες θέλουμε. Όσον αφορά ε, τα σχόλιά σας για ε, την ε, κυκλοφορία, την ελεύθερη κυκλοφορία. Συμφωνήσαμε τώρα, δεν καταλαβαίνω, με το, με το ΕΛΚ. Τώρα δεν καταλαβαίνω, κύριε Όρη, ποιο είναι το πρόβλημά σας σε αυτό το σημείο. Προβλήματα με τα συνδικάτα έχετε. Όλες οι περιπτώσεις κατάχρησης, ή τουλάχιστον αυτές που γνωρίζω εγώ, αποκαλύφθηκαν από συνδικάτα. Και εμείς στόχος μας πρέπει να είναι να προστατεύσουμε όλους τους ανθρώπους από καταχρήσεις, από εκείνους που παραβιάζουν ή δεν τηρούν τους νόμους. Επίσης, στα περισσότερα κράτη-μέλη οι έλεγχοι γίνονται και με συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων. Αυτό είναι μια πραγματικότητα και έπρεπε να τη λάβουμε υπόψη μας στην εισήγησή μας. Κοιτώντας τη Γερμανία, τον έλεγχο της μαύρης εργασίας, της αδήλωτης εργασίας, η επιθεώρηση εργασίας ελέγχει πραγματικά μόνο τις ε, συλλογικές συμβάσεις. Δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το πρόβλημα σας. Όσον αφορά τους οικιακούς εργαζόμενους, η διατύπωση συνάδει με, την, ε, με τις συμβάσεις της ΔΟΕ. Συζήτησα και με την ΔΟΕ για να διαπιστώσω αν συμφωνεί με τη διατύπωσή μου και διαπίστωσα πως ναι. Όσον αφορά την ψευτοαυτοαπασχόληση, ευχαρίστως βεβαίως ε, να συνεργαστούμε σήμερα το απόγευμα ε, πάνω σε έναν ορισμό. Τι είναι ψευτοαπασχόληση και τι είναι πραγματική αυτοαπασχόληση. Το ότι οι επιθεωρήσεις εργασίας μας θα πρέπει να ε, τύχουν συντονισμένης εκπαίδευσης το έχουμε ήδη διαπιστώσει εδώ και στις αρχές ε, του Σεπτεμβρίου. Το είπαν και οι εργοδοτικές οργανώσεις. Υπήρξαν πολλά σχόλια. Νομίζω ότι σήμερα το απόγευμα θα μπορέσουμε να βρούμε τη μία ή την άλλη λύση. Αν το ΕΛΚ δεν στηρίξει την εισήγηση αυτή, αφού θέλετε να διαγραφούν οι περισσότερες παράγραφοι, σημαίνει ότι η παρούσα κατάσταση, η ισχύουσα κατάσταση για εσάς είναι ε, ορθή, είναι ε, η ενδεδειγμένη. Αφού δεν βλέπετε την ανάγκη βελτίωσης και με αυτόν τον τρόπο, συγγνώμη, αλλά βλάπτετε και τις, ε, τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις. Ευχαριστώ. Monsieur déjà ε, εσείς μιλήσατε ήδη. Η συγγήτρια μόλις έκλεισε την συζήτηση. Μόνο εάν θέλετε να πείτε κάτι σύντομα, παρακαλώ. Αλλά συνήθως κανείς δεν είναι σύντομος. Ένα παράδειγμα θα αναδείξει το πρόβλημά μου. Ποιο είναι το πρόβλημά μου. Αυτό που θεωρώ σας παρακαλώ, σας παρακαλώ, δεν μπορώ να ξανανοίξω τη συζήτηση. Αν έχετε κάποια επιχειρήματα, μπορείτε να τα θέσετε εκτός της αιθούσης προς την εισηγήτρια. Δεν μπορώ να σας δώσω το λόγο για να κάνετε μια άλλη ανάπτυξη. Ε, θα ψηφίσουμε την πρόταση αυτή στις 26 Νοεμβρίου, αύριο δηλαδή. Ελπίζω μέχρι τότε να μπορέσουν να επιτευχθούν κι άλλες ε, συμβιβαστικές προτάσεις. Ερχόμαστε τώρα στο σημείο 5 της ημερήσιας διάταξης. Ε, θα συζητήσουμε το σχέδιο, σχέδιο έκθεσης Μαρτίν Κέσλε για, σχετικά με την έκθεση πρωτοβουλίας της Επιτροπής Γυναικών. Ε, για τις γυναίκες μετανάστριες, ε, μη νόμιμες μετανάστριες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δίνω το λόγο ε, Φου, δεν είναι εδώ ο εισηγητής. Τι να κάνω τώρα χωρίς εισηγητή. E το ΕΛΚ απουσιάζει εντελώς από αυτήν τη συνεδρίαση με την εξαίρεση δύο-τριών τώρα βουλευτών που δεν μπορούν βέβαια να πάρουν τη θέση των συναδέλφων τους. Σας δίνω το χρόνο να αυτοοργανωθείτε και περνάμε στο σημείο 6 της ημερησίας διάταξης. Αγιούντα Στάνβουρκ και πάλι για τις τροπολογίες και τις συμβιβαστικέ προτάσεις για το σχέδιο γνωμοδότησης για την Επιτροπή ΙΜΚΟ. Σχετικά με μια σχετικά με την έκθεση πρωτοβουλίας για μια ολοκληρωμένη αγορά παράδοσης δεμάτων για την ανάπτυξη ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν το ΕΛΚ βρει λύση θα επανέλθουμε στο προηγούμενο σημείο. Δίνω τώρα το λόγο στην Ιούτα Στάινρουκ για να μας παρουσιάσει τις απόψεις της για τις τροπολογίες και τις συμβιβαστικές προτάσεις που έχουν υποβληθεί μέχρι τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. 25 τροπολογίες έχουμε. Σε 6 θα ε, προσπαθούμε να βρούμε συμβιβασμούς, αλλά μετά τις τελευταίες ε, δηλώσεις. Νομίζω ότι θα καταφέρουμε να καταλήξουμε σε κοινή θέση. Επεξεργαζόμαστε ακόμα τις λεπτομέρειες βεβαίως. Ένα συμβιβασμό αφορά ε, τον έλεγχο των ορών οδήγησης και ανάπαυσης που θα πρέπει να ισχύει για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το καθεστώς τους. Ο δεύτερος συμβιβασμό αφορά την ενίσχυση ε, του ηλεκτρονικού ε, εμπορίου ως σημαντική πτυχή της ανάπτυξης. Ήταν σημαντικό και για τους κοιόδης ε, εισηγητές αυτό. Συμφωνούμε και εμείς, αλλά θα πρέπει πραγματικά να ε, εξετάσουμε ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στις ε, συνθήκες εργασίας και να εξασφαλίσουμε σωστές συνθήκες εργασίας. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν, ήταν και ο καθορισμός μέτρων μετεκπαίδευσης και τεχνικά ε, τεχνολογικές δεξιότητες, GPS για παράδειγμα. Ε, το GPS μπορεί να δώσει τόσο στους εργοδότες όσο και στους εργαζόμενους ε, να μειώσει το φόρτο, το φόρτο εργασίας τους. Και εδώ ζήτημα είναι ε, η τήρηση των συμβάσεων εργασίας, των συλλογικών συμβάσεων εργασίας στα κράτη-μέλη Επίσης πολύ σημαντική ήταν και η πληροφορία όσον αφορά τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις των επισφαλών ε, εργασιακών σχέσεων στα κοινωνικά συστήματα των κρατών μελών. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε την ε, μη παραβίαση των δικαιωμάτων των σχετικών. Έκτη, έκτος συμβιβασμός. Άνθρωποι με την ίδια εμπειρία θα πρέπει για την ίδια εργασία να λαμβάνουν την ίδια αμοιβή στον ίδιο χώρο εργασίας. Θα χαρώ πολύ να φτάσουμε σε αυτόν τον συμβιβασμό και θέλω να ευχαριστήσω όλους τους κοιόδης για την καλή συνεργασία τους. Ήμασταν χρονικά περιορισμένοι και γι' αυτό ήταν ακόμη καλύτερο το γεγονός ότι καταφέραμε και συνεργαστήκαμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κανένας από τους σκιώδεις εισηγητές δεν είναι παρόν. Είμαστε, έχουμε αργοπορήσει πάρα πολύ. Η κατάσταση εκτροχιάζεται. Θα κλείσω τη συζήτηση γιατί δεν υπάρχει και κανείς που να θέλει να πάρει το λόγο. Θα ψηφίσουμε αύριο επί του θέματος αυτού. Ο κύριος Κέσλερ, αντίθετα με αυτά που λένε, έρχεται. Θα περιμένω λοιπόν ακόμη λίγο. Ε, ερχόμαστε στο σημείο 7. Θα δώσω τον λόγο τον ε, Άνταμ Κόζακ για την έκθεση πρωτοβουλίας σε σχέση με την 7η και 8η ε, έκθεση πρόοδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την πολιτική συνοχή της ΕΕ και τη στρατηγική έκθεση του 2013 για την υλοποίηση των προγραμμάτων της περίοδου 2007-2013. Κύριε εισηγητή, έχετε το λόγο για να παρουσιάσετε τις τρεις συμβιβαστικές τροπολογίες που έχουν συνταχθεί. Έχετε το λόγο. <coughs> Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να σας παρουσιάσω τις συμβιβαστικές τροπολογίες. Επιτρέψτε μου όμως να επιφέρω μια μικρή διόρθωση. Πρόκειται για τέσσερις τροπολογίες συμβιβασμού. Έχετε δίκιο γιατί πρόκειται για τρεις συμβιβαστικές τροπολογίες συν μια άλλη τροπολογία γιατί την περασμένη εβδομάδα είχαμε μία συνάντηση με τους κοιόδης εισηγητές, ε, η οποία εκτελήχθηκε σε πολύ καλό πνεύμα και μπορέσαμε έτσι να ε, έχουμε τέσσερις αντί για τρεις ε, συμβιβαστικές λύσεις. Ε, συμβιβαστικές λύσεις που καλύπτουν 20 τροπολογίες από το ΕΛΚ, την ομάδα ΑΛΔΕ, των Σπρασίνους, τους ε, Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Ε, τροπολογίες που όλες ε, συμπεριελάμβαναν σημαντικά θέματα. Κάθε κοινοβουλευτική ομάδα συμφωνεί. Όλες οι κοινοβουλευτικές ομάδες συμφωνούν ε, με τη διόρθωση του κειμένου, ε, με την τροπολογία Β. Οι, μεγάλες, οι τέσσερις μεγάλες κοινοβουλευτικές ομάδες συμφωνούν λοιπόν επί της τροπολογίας Β. Το ίδιο μπορώ να πω και για την τροπολογία Γ. Η Δ είναι η καινούργια τροπολογία. Η τροπολογία αυτή αντικαθιστά την τροπολογία υπαριθμών 14. Ήδη είπα δεν θα έπρεπε να κατονομάσουμε συγκεκριμένες χώρες. Πρόκειται για προβλήματα που χωρίζουν τις χώρες του Βορρά και του Νότου. Το, το συμβιβαστικό κείμενο λοιπόν ε, περιλαμβάνει τα προβλήματα στα οποία αναφέρονταν, οι αρχικές τροπολογίες. Νομίζω ότι με αυτές τις τέσσερις συμβιβαστικές ε, προτάσεις μπορούμε τώρα να έχουμε μπροστά μας ένα αποδεκτό κείμενο για όλους, γιατί είναι σημαντικό να θέσουμε τον τόνο, την έμφαση ε, στην απασχόληση. Ευχαριστώ. ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Κυρία Παπαδοπούλου. Yes, thank you, Chair. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Όντω χαιρετίζουμε την έκθεση και τις προτάσεις ε, του εισηγητή του κυρίου Κώσα. Την περασμένη εβδομάδα άλλο στο Στρασβούργο καταφέραμε να βρούμε κοινό παρανομαστή για πολλές από τις συμβαστικές λύσεις, όπως είναι το σημαντικό θέμα της εγγύησης των νέων και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για όσους εγκαταλείπουν το σχολείο νωρί. Να φροντίσουμε οι μαθητές να παραμένω στο σχολείο. Επίσης, το θέμα της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης, ιδιαίτερα σε καιρούς κρίσης. Επίσης, είπαμε ότι ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στις μονογονεϊκές οικογένειες, στις πολύτεκνες οικογένειες, ε, στις οικογένειες με ανάπηρα άτομα ή με ηλικιωμένους. Χαίρομαι για τις ε, τροπολογίες μας που επικεντρώνονται σε ειδικά μέτρα για τη δημιουργία πολιτικών που θα είναι πιο φιλικές προς την οικονομική ανάπτυξη και τις βιώσιμες θέσεις απασχόλησης, γιατί οι χώρες μας ε, εφαρμόζουν πολλά μέτρα λιτότητας, ε, πολλές από τις χώρες ε, τις εφαρμόζουν και είπαμε να τις αναφέρουμε, γιατί υπάρχει μεγάλο χάσμα μεταξύ των βορείων και των νοτίων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια και οι άλλες ομάδες είναι κατά της ρητή πλειά συγκεκριμένων χωρών. Είπαμε να μην αναφέρουμε συγκεκριμένε χώρε, αλλά να αναφέρουμε το υπάρχον χάσμα μεταξύ βορείων και νοτίων χωρών τη Ευρωπαϊκή ε, Ένωση. Επειδή είπαμε επίσης να δημιουργήσουμε νέες μηχανισμούς για να καταπολεμήσουμε την ανεργία, τον κοινωνικό αποκλεισμό, να ενισχύσουμε την επιχειρηματικότητα και να αυξήσουμε τις επενδύσεις σε θέματα επιχειρηματικότητας. Τέλος, ο ρόλος των δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου θα πρέπει να επικεντρωθεί στην πρόθεση πιο ποιοτικών θέσεων εργασίας, ε, προωθώντα τη συμμετοχή ε, μειονεκτουσών μονάδων και τη δημιουργία μιας συμμετοχικής κοινωνία προσιτή σε όλου θα ήθελα να αναφέρουμε πιο ρητά το γεγονός ότι σήμερα τα μέτρα λιτότητας έχουν πολλές αρνητικές συνέπειες σε κοινωνικά θέματα και ιδιαίτερα σε κάποιες χώρες, ε, κυρίως του Νότου. Δεν καταφέραμε να συμφωνήσουμε όλες οι πολιτικές ομάδες να συμπεριλάβουμε μια πιο ισχυρή διατύπωση για το θέμα αυτό. Ελπίζω σε μια μελλοντική έκθεση να τα καταφέρουμε. Ευχαριστώ. Άλλος κανείς? Όχι. Κύριε Κόζα, θέλετε να δευτερολογήσετε. Α, και συγγνώμη, κυρία Σρέτερ. Πολύ σύντομα. Έχουμε πολύ δύσκολες διατυπώσεις στις συμβαστικές τροπολογίες, αλλά επί της αρχής, με εξαίρεση την συμβαστική πρόταση C, γάμα που δεν ξέρουμε ακόμα αν θα την υποστηρίξουμε διότι ε, δεν εμφανίζονται αυτά που θεωρούμε μη σημαντικά. Κατά τα άλλα πάντως υποστηρίζουμε τους ε, συμβιβασμούς. Στο ΣΥ, στο ΓΑΜΑ θα πρέπει να το ξαναδούμε με την πολιτική μου ομάδα αν θα μπορέσουμε να το υποστηρίξουμε αλλά όλα τα υπόλοιπα, με όλα τα υπόλοιπα δεν έχουμε καμία αντίρρηση. Ευχαριστώ. Okay. Άλλος κανείς θέλει το λόγο? Όχι. Οπότε θα ξαναδώσω το λόγο στον εισηγητή. Ευχαριστώ. Σημειώνω τι επιφυλάξει των Πρασίνων και περιμένω τις προτάσεις σα για τις συμβαστικέ ε, τροπολογίε. Κύριε Παπαδοπούλου, και εγώ προσπάθησα να συντάξω συμβαστικές τροπολογίες ε, προκειμένου να μην ικανοποιημένοι όσο το δυνατόν περισσότεροι ευρωβουλευτές και να υλοποιήσουμε τους στόχους μας. Γιατί μην ξεχνάτε ότι το κείμενο δεν είναι νομοθετικό. Πρόκειται για μια διαδικασία που ξεκίνησε από την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης και εμείς θέλουμε να εστιάσουμε την προσοχή μας σε τομείς για τους οποίους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αργότερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορούν να παρέμβουν. Και θα πρέπει να επιστήσουν την προσοχή τους στους τομείς αυτούς για να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες. Μια και πρόκειται λοιπόν για μη νομοθετική έκθεση, πολύ σπάνια α, καταλήγει σε συγκεκριμένες νομοθετικές προτάσεις. Απλώς εφιστά την προσοχή των διαφόρων πλευρών σε συγκεκριμένα θέματα. Και Ελπίζω αύριο να εγκρίνουμε την γνωμοδότηση και να λάβει υπόψη τις προτάσεις μας και η αρμόδια επιτροπή καθήλη. Λαμπρά, ολοκληρώσαμε και το σημείο 7. Θα ψηφίσουμε την γνωμοδότηση του κυρίου Κώσα αύριο το πρωί. Στο μεταξύ έφτασε και ο κύριος Κάστλερ. με 40, 40 λεπτή καθυστέρηση. Επανερχόμαστε λοιπόν στο σημείο 5 της της διάταξης. Θα δώσω το λόγο στο συντάκτη γνωμοδότησης για να μας παρουσιάσει τις 5 συμβαστικές τροπολογίες ε, στη γνωμοδότηση που έχει θέμα τις μετανάστριες που δεν διαθέτουν επίσημα έγγραφα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για γνωμοδότηση που θα δώσουμε στην κατ' ουσίαν αρμόδια επιτροπή, την Επιτροπή Γυναικών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς να ευχαριστήσω όλους τους κυριώδεις συζητητές. Νομίζω ότι είχαμε μια καλή συνεργασία στον τομέα των μεταναστριών που δεν διαθέτουν επίσημα έγγραφα και καταφέραμε να επιτύχουμε να παρουσιάσουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα εισήγηση. Νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε στους συμβιβασμούς. Σε κάποιους τομείς είχαμε κάποιες δυσκολίες, θα το πω ανοιχτά διότι στην εισήγηση αυτή θεωρώ σημαντικό να αναφερθούμε και σε συγκεκριμένα προβλήματα που σχετίζονται με παιδιά, εγκυμοσύνες. Σε, αυτήν την, σε αυτό το ζήτημα θα υπάρχει μια τροπολογία που εγώ δεν ε, υποστηρίζω Σε αυτό το ένα σημείο λοιπόν, παρότι έχω διαφορετική θέση, ελπίζω στην ψηφοφορία να καταλήξουμε σε καλό τέλος, αλλά θέλω να το τονίσω ε, ότι εγώ έχω άλλη γνώμη. Νομίζω ότι θα μπορέσουμε να ε, είμαστε όλοι ικανοποιημένοι με τους συμβιβασμούς και νομίζω ότι θα μπορέσει να έχει θετικές επιπτώσεις και για την Επιτροπή Γυναικών η συγκεκριμένη εισήγησή μου. Ευχαριστώ. Η κυρία Γιακονσάρη. Yhteistyöstä Martin Kastlerille oli tietenkin... Ευχαριστώ για τη συνεργασία με τον Μάρτιν Κάσλερ. Βεβαίως ήταν λίγο έκπληξη Ε το ότι είπατε ότι μία, ένας σημαντικός συμβιβασμός ε, δεν μπορεί να τύχει της ε, υποστήριξής σας. Δεν το καταλαβαίνω, διότι τα γέννητα παιδιά, η προστασία αυτών των παιδιών προϋποθέτει βεβαίως και την προστασία των εγγύων. Και υπάρχει ένα κόκκινο νήμα που συνδέει τα ζητήματα αυτά, που είναι η υγεία των γυναικών και η προστασία των εγγύων. Με αυτόν τον τρόπο ε, μπορούμε να προστατεύσουμε και τα παιδιά και νομίζω ότι είναι βασικό το ερώτημα αυτό πρέπει να μας ενδιαφέρει και αυτό το ζήτημα, διότι όταν εξετάζουμε ποιες ομάδες στην Ευρώπη βρίσκονται στην ε, δυσχερέστερη θέση, ε, τότε είναι ακριβώς οι γυναίκες που δεν διαθέτουν επίσημα έγγραφα. Γι' αυτό είναι σημαντικό οι γυναίκες αυτές να έχουν ίση μεταχείριση, να έχουν πρόσβαση στην υγεία, να έχουν τη δυνατότητα να εργάζονται και να ε, μπορούν να ζήσουν αυτόνομα δεν επιτρέπεται να ε, τις μεταχειρίζεται κανείς ως σκλάβες, ως δούλες που δυστυχώς είναι μια πραγματικότητα, μια, μια μεγάλη ντροπή για την Ευρώπη. Κατά τα άλλα να σας ευχαριστήσω για τη συνεργασία βεβαίως. Ε, μια παρατήρηση επίσης. Βλέπω εδώ ότι το γραφείο μετάφρασης χρησιμοποιεί τον όρο παράνομοι μετανάστες. Οι άνθρωποι δεν είναι παράνομοι. Στα φινλανδικά υπάρχει ο όρος για τους ανθρώπους που δεν διαθέτουν έγγραφα. Ναι, αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστώ. Τέλεια. Θέλει κάποιος άλλος να λάβει το λόγο. Δεν βλέπω κάποιον. Κύριε Κάστλερ, θέλετε να απαντήσετε. Όχι. Θα το κάνετε σε διμερή βάση, υποθέτω. Ολοκληρώσαμε λοιπόν και το σημείο αυτό. Αύριο θα ψηφίσουμε κατά τη διάρκεια του χρόνου που είναι αφιερωμένο στις ψηφοφορίες. Για το σημείο 8 θα εξετάσουμε τη συνεισφορά μας στο ε, έργο της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων για για τη βελτίωση της καταλληλότητας και της αποδοτικότητας του κανονιστικού πλαισίου. REFIT, αποτελέσματα και επόμενα βήματα. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και όπως ξέρετε, κατά τη διάσκεψη των Προέδρων της Επιτροπής ε, συμφωνήθηκε κάθε κοινοβουλευτική επιτροπή ε, η οποία ενέχεται στην, στον κατάλογο προτάσεων που εμπίπτουν στην ανακοίνωση REFIT της Δευτέρας Οκτωβρίου 2013 ε, θα συμνισφέρει στο σχέδιο ψηφίσματος. Έτσι λοιπόν και η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων θα συνεισφέρει. Ε, ήταν μικρή η προθεσμία, ήταν σύντομη η προθεσμία για τις τροπολογίες, κατά αποτέλεσμα 19 τροπολογίες, 4, 4 από την ομάδα ECR, μία από την ομάδα των Πρασίνων, με τις ίδιες προϋποθέσεις, ε, χωρίς ε, να λαμβάνει υπόψη το σχέδιο ψηφίσματος της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων. 14 τροπολογίες για το σχέδιο ψηφίσματος της Επιτροπής αυτής. Ε, από την πλευρά μου, βλέποντας την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων, και του εισηγητή, του κυρίου Καρίμα, ε, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να ακουστεί η φωνή της Επιτροπής μας. Γιατί όπως ξέρετε η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, ήταν πολύ σκληρή ε, σε σχέση με τις αρμοδιότητές μας. Δεν έλαβε απόψη της, της, τη συμφωνία μεταξύ των κοινωνικών εταίρων Ε, και σε σχέση με τις ε, μειοσκελετικές διαταραχές, ένα θέμα που εδώ και πολύ καιρό μας απασχολεί ε, και πάλι και αυτό έμεινε εκτός. Θα, νομίζω ότι πρέπει να στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα στη Νομική Επιτροπή. Αυτά τα λίγα είχα να πω. Και από αυτήν την άποψη κάποιες τροπολογίες που υπέβαλε η ομάδα ESR, ECR, ίσως παρουσιάζει κάποια προβλήματα, συγκεκριμένα η 14, η οποία ε, θεωρεί ότι η οδηγία είναι πολύπλοκη, δεν ε, είναι καθόλου ευέλικτη και είναι πολύ, πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ε, αν δούμε τα, τη στάση που είχε τηρήσει η Επιτροπή τελευταίως, δυσκολευόμαστε να καταλάβουμε αυτή την άποψη. Στη ΔΕΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 19 ε, γίνεται λόγος για τους κοινωνικούς εταίρους ε, όταν οι ίδιοι κοινωνικοί εταίροι κάνουν κάποια μελέτη αντικτύπου. Δεν ξέρω αν μπορούμε να ζητήσουμε κάτι τέτοιο με ένα τέτοιο κείμενο να δώσουμε μια, πολύ, μια νέα διάσταση, πολύ πιο περίπλοκη στον τρόπο λειτουργίας των ε, κοινών συμφωνιών, των κοινωνικών εταίρων. Δεν... Θα ήθελα να δώσω τον λόγο στην κυρία Γκρίνμπεργκ. Καταρχήν θέλει και κάποιος άλλος να λάβει το λόγο, ο Τσαβάουρη και η Ελίζαμπεθ Σρέντερ στη συνέχεια. Αυτούς τους τρεις ομιλητές λοιπόν θα ακούσουμε. Η Εύελιν Ρέντνερ καταρχήν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρόκειται για θεμελιώδεις, ε, θεμελιώδη θέματα. Θα μιλήσω αμέσως, ευθύς αμέσως για τις τροπολογίες της ομάδας ECR. Ε, υπάρχει κάτι που θα ήθελα να αμφισβητήσω και συγκεκριμένα την άποψη ότι πρέπει να πηγαίνουμε πάντοτε για το maximum. Πρόκειται για ένα σύστημα που διατράνωσε ο Ζακ Ντελόρ, ένα σύστημα σύμφωνα με το οποίο οι κοινωνικοί εταίροι πρέπει να ενισχυθούν μέσω του τομεακού ε, διαλόγου και μέσω διατομεακών συμφωνιών. Συμφωνιών δηλαδή εγκάρσεων σε πολλούς τομείς. Δεν νομίζω ότι καταστρέφοντας ολοσχερός το σύστημα αυτό είναι ο σωστός τρόπος για να προχωρήσουμε. Ε, για μένα αυτό είναι πάρα πολύ σαφές. Δεν πρέπει να αμφισβητηθεί το σύστημα αυτό. Περί τίνος πρόκειται. Πρόκειται για την ε, συμφωνία των κομωτών, για παράδειγμα και θεωρούμε ότι μπορεί να λυθεί το πρόβλημα σε, στο, σε τομεακό επίπεδο. Ωστόσο, αυτό θα λυθεί υπόψη για μια σειρά άλλων θεμάτων. Έχουμε το θέμα του κοινωνικού διαλόγου που υπερβαίνει τους τομείς. Πρέπει κατά τη γνώμη μου να είμαστε πάρα πολύ σαφείς το refit και μιλώ για τις δικές μου τροπολογίες όσο αφορά την ασφάλεια και την υγιεινή. Τα θέματα αυτά δεν πρέπει να υπονομευθούν. Το ίδιο ισχύει και με την προστασία των καταναλωτών. Και τι συμβαίνει εδώ. Θα πρέπει να μειώσουμε και τα βάρη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά όχι σε βάρος της προστασίας των εργαζομένων ή της υγιεινής και της ασφάλειας στους χώρους εργασίας το επιχείρημα αυτό πρέπει να το τονίσουμε, γιατί οι ίδιες οι κοινωνικές συμφωνίες, οι ίδιοι κοινωνικοί εταίροι μέσω των συμφωνητών τους συμβάλλουν στην ευρωπαϊκή νομοθεσία εν τέλει. Όλη λοιπόν η διαδικασία που προτείνεται από το ECR είναι να γίνεται μία ανεξάρτητη ξεχωριστή μελέτη αντικτύπου. Αυτό απορρίφθηκε γιατί ε, δήθεν θα υπονόμευε την ε, ε, οικονομική κατάσταση στην Ευρώπη. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να ενισχύουμε τους κοινωνικούς εταίρους, όχι να τους αποδυναμώνουμε και πρέπει να σκεφτούμε και την πίεση υπό την οποία τελούν οι κοινωνικοί εταίροι αυτή τη στιγμή στο πλαίσιο αυτής της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης. Οι κοινωνικοί εταίροι αποδυναμώνονται αυτή την περίοδο, δεν ενισχύονται. Και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις επίσης θα πρέπει αυτά τα πράγματα να ισχύουν μόνο να δικαιολογούνται σε κοινωνικό επίπεδο. Ένα πολύ σαφές μήνυμα λοιπόν. Οι κοινωνικοί εταίροι, οι συμφωνίες μεταξύ των κοινωνικών εταίρων πρέπει να τεθούν σε άμεση εφαρμογή, πρέπει να τίθενται γενικά σε άμεση εφαρμογή χωρίς ε, να προσπαθούμε ε, να βρούμε εναλλακτικέ μεθοδεύσει για να παρακάμψουμε τις συμφωνίες των κοινωνικών εταίρων, πράγμα που συμβαίνει σε πάρα πολλές φορές. Ευχαριστώ κύριο Σόρη και μετά κύριο Σιρότερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Διάβασα την έκθεση και συμφωνώ με το περιεχόμενό της. Γι' αυτό μάλιστα και δεν κατέθεσε ούτε καν τροπολογίες, γιατί στενίζομαι πλήρως το περιεχόμενο της έκθεσης. Διάβασα τις υπόλοιπες τροπολογίες, με μερικές συμφωνώ, με άλλες διαφωνώ. Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά την οδηγία για την εργασία και τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Η ομάδα συντηρητικών και μεταρρυθμιστών ε, έχει γνώμη με την οποία δεν συμφωνούμε. Επαναλαμβάνω, δεν συμφωνώ με όλες τις τροπολογίες. Αλλά με το κείμενο δεν έχω πρόβλημα. Πιστεύω ότι είναι σωστό και αν γίνεται θα επιθυμούσα να ελαφρύνουμε το γραφειοκρατικό άχθος και να περιοριστούμε στα ουσιώδη για να είναι πιο εύκολη και εφαρμογή των ε, νομοθετικών διατάξεων. Σε ό,τι αφορά τις προτάσεις των μεταρρυθμιστών και συντηρητικών, αυτή τη φορά δεν μπορούμε να τις ε, υποστηρίξουμε όπως κάνουμε άλλες φορές. Ευχαριστώ. Η κυρία Σρέτερ. Ευχαριστώ. Φυσικά αυτό που με ενδιαφέρει είναι η εισηγήτρια αν θα δεχτεί τις τροπολογίες μας. Έχω ένα πρόβλημα με το πρόγραμμα που αφορά την προστασία των εργαζομένων. γιατί φαίνεται να υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα προστασίας της εργασίας. Οπότε ε, οι μεγάλες επιχειρήσεις υποχρεούνται να προστατεύσουν τους εργαζόμενους τους, ενώ κάτι τέτοιο δεν ισχύει για τις μικρομεσαίες. Δεν νομίζω ότι είναι αυτός ο στόχος μας, γιατί η υγεία και προστασία ε, και ασφάλεια των εργαζομένων είναι οικουμενικές αρχές. Δεν θα πρέπει να υπάρχει διαφορά από τη στιγμή που μιλούμε για την ίδια εργασία δεν θα πρέπει να υπάρχει διαφορά ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης. Εδώ έχουμε ευρωπαϊκούς κανόνες και δεν θα πρέπει αυτοί οι κανόνες να θεσπίζουν διακρίσεις. Πιστεύω ότι στην περίπτωση αυτή η κοινοτική νομοθεσία δεν είναι υπερβολικά σχολαστική και και ούτε είναι υπερβολική η κοινοτική ρυθμίση σε θέματα αυτά. Δεν μπορούμε όμως να κάνουμε διακρίσει μεταξύ της προστασίας του εργαζόμενου ανάλογα με το αν η επιχείρηση στην οποία απασχολείται είναι μεγάλη ή μικρή. Το θέμα της υγείας και της ασφάλειας και ο σεβασμός της υγείας και της ασφάλειας η προστασία τους είναι ένα αναφέρετο δικαίωμα που κατοχυρώνεται από την ίδια τη συνθήκη. Θα πρέπει λοιπόν η υποχρέωση προστασία να βαρύνει όλε τι επιχειρήσει άσχετα με το μέγεθό του. Πολύ σημαντικό αυτό το θέμα και ελπίζω να συμφωνήσει μαζί μα η συγκεκριά. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σέρκας. Ευχαριστώ. Θα ήθελα, κυρία Πρόεδρε, να πω ότι η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Και εδώ μιλούμε για μια έκθεση που για τους σοσιαλιστές έχει ιδιαίτερη σημασία σε μια στιγμή πολύ χαλεπή εξαιτία της ε, πολύ σοβαρή χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση και ακόμη σοβαρότερη κοινωνική κρίση, για να μην μιλήσω για την πολιτική κρίση στην Ευρώπη. Οπότε, αν συνεχίσουμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αλλού με προγράμματα που αντί να δίνουν ασφάλεια στους πολίτες, ε, που αντί να προστατεύουμε τη ζωή τους, ε, τα θεμελιώδη τους δικαιώματα, ουσιαστικά παλιδρομούμε σε σχέση με ήδη κεκτημένα δικαιώματα και προδιαγραφέ, αυτή η αδιαφορία των Ευρωπαίων πολιτών απέναντι στην Ένωση και η απομάκρυνσή του θα αυξηθεί. Γιατί υπάρχουν κάποιοι που δεν θα έλεγα ότι είναι εχθροί της Ευρώπης, αλλά υπάρχουν ομάδες που θέλουν ε, η Ευρώπη να οικοδομηθεί σε πάγιες ε, και οικουμενικέ αξίες. Και έχουμε πέσει σε μια παγίδα, γιατί μιλούμε για το εύνομο θετήν, ενώ ε, μερικές ομάδες θέλουν την πλήρη απελευθέρωση και την κατάργηση οποιασδήποτε ρύθμιση. Έτσι όμως θα γράψουν ένα ακόμη κεφάλαιο στην καταστροφή α, του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Γιατί δεν αξίζει ε, να παίρνουμε ένα λευκό χαρτί και να γράφει ο καθένας ό,τι του κατέβει στο κεφάλι. Εδώ έχουμε μια ιστορία, έχουμε συνθήκες, έχουμε χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων, έχουμε ένα Συμβούλιο της Ευρώπης με συγκεκριμένες συμβάσεις τις οποίες έχει προσυπογράψει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε συμβάσει τη ΔΟΕ, Τη διεθνή οργάνωση εργασία. Δεν μπορούμε να κάνουμε τάμπουλα ράσα και μόνο υπό το πρόσχημα της ε, κατάργηση γραφειοκρατικών διατυπώσεων να καταπατάμε τα κεκτημένα δικαιώματα των εργαζομένων. Ε, μπορούμε να κάνουμε πιο ελαστική την νομοθεσία, μπορούμε να άρουμε τα εμπόδια στην απρόσκοπτη επιχείρηση των ε, επιχειρήσεων, αλλά είμαστε αμετάβλητοι, αμετακίνητοι και αδιάλεκτοι ε, και είμαστε κατά των παλινδρομήσεων και της καταπάτησης των κεκτημένων. Δεν μπορούμε να θυσιάζουμε εδώ ένα θεμελιώδης δικαίωμα που είναι η ασφάλεια των εργαζομένων και η προστασία τους σε περίπτωση ασθένειας, σε περίπτωση εργασιακού ατυχήματο. Σε καμία περίπτωση δεν θα ασθενιστούμε ε, μια τέτοια πρόταση αν ακολουθήσει αυτή την ιδεολογική γραμμή. Και θα ζητούσα από τους συναδέλφους των άλλων πολιτικών ομάδων να σκεφτούν το θέμα πολύ σοβαρά, γιατί οι προκλήσεις είναι σοβαρές και εμφανίζονται σε όλες τις χώρες. Αν θέλετε να γεμίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με εξτρεμιστέ, με ακροδεξιού ή ακροαριστερού και ευρωσκεπτικιστέ, εντάξει, αυτό να κάνουμε. Να καταστρέψουμε τον κοινωνικό διάλογο, να καταστρέψουμε την κοινωτική νομοθεσία. Αλλά εδώ μιλούμε για δύο πυλώνε τη κοινωνική Ευρώπη και δύο βασικού πυλώνε τη ευρωπαϊκή ηθαγένεια. Ευχαριστώ. Merci. ευχαριστώ. Αύριο θα γίνει ψηφοφορία για το θέμα αυτό. Δεν έχω άλλα σχόλια. Πάντως ε, εκπλήσωμε που στις τροπολογίες που έχουν υποβληθεί, όταν βλέπουμε το πεδίο που καλύπτει η ανακοίνωση της Δευτέρας Οκτωβρίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διαπιστώνουμε ότι το θέμα της οδηγίας για τις ε, μυοσκελετικές διαταραχές που ζητούσαμε και περιμέναμε καθ' τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής αιτίας έχει αποσυρθεί. Πραγματικά κρίμα. Με θλίβει ιδιαίτερα αυτή η παράληψη. Έπρεπε να είχα ασχοληθεί προσωπικά με το θέμα αυτό. Θα ψηφίσουμε, επαναλαμβάνω, αύριο τις τροπολογίες και ελπίζω να στείλουμε ένα καλό μήνυμα στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Ολοκληρώσαμε το σημείο 8 και περνάμε στο σημείο 9. Θα δώσω το λόγο στο Σέρχιο Γκουτιέρες, Πριέτο, για να μας παρουσιάσει την γνωμοδότησή του και τις 30 τροπολογίες που έχουν υποβληθεί για την γνωμοδότησή του με θέμα την μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής οικονομίας. Γνωμοδότηση που θα εγχειρήσουμε στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων. Κύριε Σιγητά, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω ειλικρινά τους συναδέλφους για τη συνεργασία τους και για τις τροπολογίες τους που συμπληρώνουν, βελτιώνουν και διορθώνουν ε, μερικές παραγράφους της γνωμοδότησής μου. Ελπίζω να καταλήξουμε στη συμβαστική λύση. Ανεξάρτητα όμως με τις συμβαστικές προτάσεις θα ήθελα να επισημάνω κάποιες ιδέες που είναι κατά τη γνώμη μου πολύ σημαντικές και υποβλήθηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Καταρχήν, για να δημιουργήσουμε ένα πρόσφορο έδαφος για τις ε, μακροπρόθεσμες μας ε, προτάσεις, όπως φαίνεται και από τη γνωμοδότηση και από τις τροπολογίες, θα πρέπει να αυξήσουμε τη σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών ε, αγορών και τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση. Έτσι θα μειώσουμε και το κόστος των επιχειρήσεων και θα βελτιώσουμε τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Ταυτόχρονα πιστεύουμε ότι ακριβώς επειδή είμαστε υπέρ της μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης στη χρηματοδότηση, αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε αναφαδόν κατά της βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης. Αντίθετα, θεωρούμε ότι θα πρέπει να υποστηρίξουμε και τη βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση. Αλλά επενδύοντας τη μακροπρόθεσμη προοπτική θα διορθώσουμε μερικά από τα κακά τα δεινά των τελευταίων ε, καιρών που ακριβώς εξαιτίας της βραχυπρόθεσμης συμπεριφοράς στις χρηματοπιστωτικές αγορές ε, ενισχύσαμε την ε, κερδοσκοπική οικονομία εις βάρος της παραγωγικής και της πραγματικής οικονομίας. Θεωρούμε λοιπόν ότι τέτοιου είδους μακροπρόθεσμες επενδύσεις εξασφαλίζουν πολύ μεγαλύτερη σταθερότητα. Γι' αυτό τις υποστηρίζουμε και πιστεύω ότι με υπεύθυνε δημόσιες αρχές λογικό είναι να περιμένουμε μια τέτοια συμπεριφορά και μία πρόθεση της ε, μακροπρόθεσμας ε, προοπτικής. Η κυρία Καστές στην τροπολογία της ε, μας υπεθυμίζει τις μέσοπρόθεσμες δεσμεύσεις μας ό,τι αφορά την ψηφιακή, ψηφιοποίηση, την ενέργεια και θεωρεί η κυρία Καστέξη στην τροπολογία 12 ότι αυτές οι προτεραιότητες θα πρέπει να αποτελούν κοινωνικές προτεραιότητες ώστε οι νέοι μηχανισμοί χρηματοδότησης και οι σχετικέ διευκολύνσει που γίνονται από τι δημόσιε αρχέ θα πρέπει να προσανατολίζονται σε τέτοιου είδου επενδύσει. Επίση, προσθέτει μία παράγραφο πολύ σημαντική που ζητά περισσότερες κοινοτικέ αρμοδιότητε ώστε να μην αναχαιτιστούν τέτοιε επενδύσει ή να μην δοθούν αντικίνητρα για τέτοιε επενδύσει. Κάτι πολύ σημαντικό είναι οι τροπολογίε που βελτιώνουν τι προτάσει μου σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση, την έλλειψη πρόσβαση στη χρηματοδότηση που ταλανίζει τι μικρομεσαίε επιχειρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι μόνο εξαιτία των διαφορών που υπάρχουν σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στην παραδοσιακή πίστη εκ μέρου των ε, μικρομεσαίων επιχειρήσεων, υπάρχουν διαφορέ 4-6% μεταξύ των κρατών μελών, αλλά επειδή στην πράξη ουσιαστικά οι μικρομεσαίε επιχειρήσει δεν έχουν καν πρόσβαση σε εναλλακτικά συστήματα χρηματοδότηση των, ε, του κεφαλαίου χρησιμοποιείται από τις, από, τους μεγάλες, ε, από τους μεγάλους ομίλους και τις πολυεθνικές εταιρείε. Υπάρχουν τεράστιες διαφορές σε ό,τι αφορά τις μακροπρόθεσμες χρηματοδοτήσεις μεταξύ μικρών και μεγάλων ε, εταιριών και χαιρετίζουμε τις τροπολογίες που προτείνουν ή απαιτούν λύσεις του προβλήματος αυτού. Θεωρώ ότι για να μειώσουμε την εξάρτηση που έχουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις από τον τραπεζικό τομέα, το 70% της χρηματοδότησής τους εξαρτάται ή προέρχεται από το παραδοσιακό σύστημα δανεισμού, το 70% είναι υπερβολικό ποσοστό, θα πρέπει να το μειώσουμε και να μειώσουμε αυτή την εξάρτηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από τις τράπεζες. Και επίσης θεωρούμε ότι οι μηχανισμοί χρηματοδότησης θα πρέπει να εξυπηρετούν ε, και την αναχρηματοδότηση του συστήματος ε, και όχι μόνο την εξυπηρέτηση των ε, παλιών υποχρεώσεων. Επίσης θέλουμε καλύτερο συντονισμό των ε, κοινοτικών διατάξεων και την, το τρόπο εφαρμογής του στα διάφορα κράτη-μέλη. Θα πρέπει να βρει τρόπους η Ευρωπαϊκή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να προωθήσει το καλύτερο συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών στα θέματα αυτά. Πιστεύω ότι έχουμε ήδη μια καλή βάση για να διαμορφώσουμε μια ωραία έκθεση και επαναλαμβάνω οι τρο, πολλές τροπολογίες επισημαίνουν σημαντικές προτεραιότητες που με βρίσκουν σύμφωνο και πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε ευρεία συνένεση για το περιεχόμενο της γραμματότησης πριν περάσουμε στην ψηφοφορία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. κυρία Σάια, που αν δεν κάνω λάθος, αντικαθιστά το σκιώδη εισηγητή του ΕΛΚ, τον κύριο Και μετά ο Φιλίπ Μπέινον. Ευχαριστώ. Εκ μέρους του κύριου Ουγγουρ, θα ήθελα να σας πω ε, τη γνώμη του για το θέμα αυτό. Θα ήθελε πρώτα απ' όλα να τονίσει ορισμένε πτυχές που αφορούν στις τροπολογίες όσον αφορά τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση. Η γνωμοδότηση αυτή είναι από τις σημαντικότερες με τις οποίες έχουμε ασχοληθεί την τελευταία περίοδο. Για να προσεγγίσουμε σωστά το ζήτημα ε, της οικονομικής ανάπτυξης είναι σημαντικό να συμφωνήσουμε σε μια στρατηγική που θα οδηγήσει στην οικονομική ε, ανάκαμψη. Από τις 13 τροπολογίες παρατηρεί ο σκιώδης εξωτικής ότι πολλά σχετίζονται με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, την ανάπτυξη ενός ε, συστήματος χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αναπτυξιακές τράπεζες ώστε να αυξήσουν τη χρηματοδότησή τους και τη η γεφύρωση των εθνικών στρατηγικών με την μακροπρόθεση στρατηγική. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά ζητήματα όσον αφορά το θέμα που συζητούμε. Όσον αφορά για την προστασία των εργαζομένων θα πρέπει να δημιουργήσουμε το περιβάλλον για την εξέβρεση εργασίας που είναι σημαντικό για την επανέναρξη των οικονομικών δραστηριοτήτων, για την ανάπτυξη, την ανάκαμψη. Πολλές από τις τροπολογίες αφορούν στο ίδιο αυτό θέμα. Και γι' αυτό το λόγο θεωρεί ότι εύκολα θα καταλήξουμε, στην, ε, ε, θα καταλήξουμε σε συμβιβασμό. Ευχαριστώ. Αυτά ήθελα να πει ο Σκιώδης Συγητής. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι το σχέδιο γνωμοδότησης είναι περιεκτικό. Ε, γι' αυτό και ε, υπέβαλα κάποιες μόνο τροπολογίες. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να επικεντρώσουμε στις, ε, στα πλεονεκτήματα της μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης και όχι στα μειονεκτήματα της βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης. Επίσης, υπάρχουν πολλές απόψεις από τις οποίες μια μακροπρόθεσμη στρατηγική βοηθά και τους επενδυτές και η μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση είναι μόνο μία πτυχή στην παράγραφο 2 νομίζω ότι είναι καλύτερα να εστιάσουμε στους στόχους που η μακροπρόθεσμη ε, χρηματοδότηση θα πρέπει να επιδιώκει. Επίσης θεωρώ ότι είναι σωστό να, να τονίσουμε το ρόλο των καινοτόμων μορφών χρηματοδότησης ώστε εργαζόμενοι, καταναλωτές και πολίτες να επωφελούνται. Στην παράγραφο 3 προτείνω τροπολογία για την εξαίρεση, για τη διαγραφή της αναφοράς στην κτηματομεσητική αγορά, ανταλαμβάνομαι την ισπανική οπτική του εισηγητή, αλλά παρόλα αυτά πιστεύω ότι και σε αυτόν τον τομέα στον, ε, της αγορά αγοράς υπάρχει προοπτική δημιουργίας θέσεων απασχόλησης στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό δεν νομίζω ότι είναι σωστό να πούμε ότι η κτηματομεσιστική αγορά δεν μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη. Οπότε δεν νομίζω ότι θα πρέπει να εξαιρείται από τα μελλοντικά χρηματοδοτικά προγράμματα. Τέλος, θα ήθελα να ενισχυθεί η παράγραφος 4 μέσω της απλοποίησης της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση. Και το συζητήσαμε αυτό και με τον εισηγητή και νομίζω ότι συμφωνεί μαζί μου. Ευχαριστώ. Θέλουν άλλοι να λάβουν το λόγο. Αν όχι, νομίζω ότι πρέπει να ε, συζητήσετε με τον εισηγητή, να ανταλλάξετε απόψεις. Τέλος πάντων, θέλει κάποιος άλλος να λάβει το λόγο. Όχι. Ίσως λοιπόν ο εισηγητής, ο εισηγητής θέλει να ξαναλάβει το λόγο. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Απλώς θα ήθελα να ευχαριστήσω τους δύο συναδέλφους που πήραν το λόγο. Να πω ότι κατά βάση συμφωνούμε, όπως είπαν και οι προλαλήσαντες. Και είναι σημαντικό, όπως είπε η κυρία Σάια, να βρούμε χρηματοδότηση πέραν των τραπεζών. Γιατί ούτως ή άλλως ε, οι επιχειρήσεις δεν έχουν πια πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό. Και όπως είπε ο κύριος Μπένιον, θα πρέπει να είμαστε φάνταστοι και ευρηματικοί, να βρούμε νέους μηχανισμούς που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση μερικές φορές ήδη και δεν χρησιμοποιούνται. Να επωφεληθούμε και από τις εμπειρίες άλλων οικονομικών εταίρων μας. Τώρα για τον κτηματομεσητικό κλάδο έχουμε κάποιες διαφορές. Όντως, ε, στην Ισπανία είχαμε αυτή τη φούσκα ε, στα, στα ακίνητα, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι μόνο ισπανικό το πρόβλημα. Αντίστοιχα φαινόμενα είχαμε όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε άλλες χώρες, αλλά και σε άλλες περιοχές του κόσμου. Και γινόταν η εξαίρεση του τομέα των ακινήτων, δίνοντας έμφαση στις, ε, στην κοινωνική αιστεία, στις, στις εργατικές κατοικίες, για να αντιμετωπιστούν ε, ιδιαίτερα οι αρνητικές συνέπειες της φούσκας ε, στα, των ακινήτων. Πάντως ήταν πολύ επικοδομητικές οι τροπολογίες του κυρίου Μπένιον ε, και συμφωνώ, τουλάχιστον με συντριπτική πλειοψηφία των σημείων του. Ευχαριστώ και πάλι τους συναδέλφους που πήραν το λόγο και ευχαριστώ για τις τροπολογίες τους που βελτιώνουν αισθητά τις δικές μου προτάσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ψηφίσουμε Στις 5 Δεκεμβρίου οι συμβιβαστικές τροπολογίες. Στις 9 θα ψηφίσουμε επί της γνωμοδότησης. Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή θα αποφανθεί στις 20 Ιανουαρίου. Ολοκληρώσαμε και αυτό το σημείο. Περνάμε στο σημείο 10 της ημερησίας διάταξης. Ξαναδίνω το λόγο στον κύριο Μάρτιν Κάστλερ για να παρουσιάσει τις 27 τροπολογίες που κατατέθηκαν για το σχέδιο γνωμοδότησης ε, σχετικά με την Επιτροπή ΙΜΚΟ για το Solvit, κύριε Σιγητά, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι θα είμαι πολύ σύντομος. Να ευχαριστήσω για τις 27 τροπολογίες αυτά θα μπορούσε ίσως να δημιουργηθεί κάποια σύγκρουση, να αναφέρω στις τρεις μεγάλες ομάδες. Μιλούμε για τους ε, μετακινούμενους εργαζόμενους και τα προβλήματά τους εντός της ενίας αγοράς. Αφετέρου ε, μιλούμε για τους ανθρώπους με περιορισμούς μέσω του Solvit και μέσω της πρόσβασης στην ιστοσελίδα της Solvit και τρίτο θέμα αφορά πάλι τους ε, μετακινούμενους ε, εργαζόμενους πώς θα μπορέσουμε στον τομέα των συντάξεων και, των, ε, και της κοινωνικής ασφάλισης να τους υποστηρίξουμε νομίζω ότι το εργαλείο αυτό το Solvit είναι άγνωστο εν πολλής δεν χρησιμοποιείται επαρκώς το ε, τόνισαν και αυτό και άλλοι συνάδελφοι και θέλω να συμφωνήσω και εγώ με αυτό ότι ε, ενδεχομένως ε, χρειαζόμαστε και μια κάποια αύξηση των, ε, των δημοσίων σχέσεων. Ένας συνάδελφος πρότεινε να ενσωματωθεί το Solvit σε αυτό το ευρωπαϊκό έτος πολιτών. Από αυτή την άποψη νομίζω ότι 27 τροπολογίες αφορούν τρεις-τέσσερις μεγάλους συμβιβασμούς και ελπίζω να καταφέρουμε να καταλήξουμε σε μια καλή λύση. Γενικά να πω ότι με την γνωμοδότησή μας αυτή θέλουμε για άλλη μια φορά να διαφημίσουμε το εργαλείο αυτό, το Solvit, και να καλέσουμε ε, για τη χρήση τους, ιδιαίτερα στον τομέα των ε, των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν. Ε, σκέφτομαι και την, ε, ε, μια παλαιότερη γνωμοδότηση όσον αφορά το dumping. Κάποια από αυτά τα ζητήματα μπορούν να αποτυπωθούν καλύτερα και μέσω του Solvit και γι' αυτόν τον λόγο θα χαιρόμουν ιδιαίτερα αν καταφέρουμε να καταλήξουμε σε αυτή τη συμβαστική λύση ώστε να μπορέσουμε να διαφημίσουμε περαιτέρω το Solvit, ώστε οι πολίτες να μην προσφεύγουν στα δικαστήρια κατευθείαν αλλά να μπορέσουμε χωρίς μεγάλο κόστος να τους προσφέρουμε υποστήριξη μέσω τέτοιων δικτύων. Ευχαριστώ πολύ. Θέλει κάποιος να λάβει το λόγο. Παρακαλώ, η κυρία Μπαλντακίνο. Άλλος κάποιος θέλει να λάβει το λόγο, ο κύριος Μπεντένιον. Όχι, ο κύριος Μπένιον. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Όπως ε, είπε και ο εισηγητής, ε, μπορούμε να υποστηρίξουμε την πλειοψηφία των ε, τροπολογιών που έχουν υποβληθεί. Πολλές τροπολογίες αυξάνουν την ορατότητα των δικτύων Solvit τόσο στο διαδίκτυο μέσω διασύνδεσης με άλλες ε, πύλες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, μεταξύ συμβουλευτικών επιτροπών, ε, αρχών, φορέων, αρμόδιων για τα κοινωνικά συστήματα. Και για τους πολίτες όμως, για να είμαστε πιο κοντά στους πολίτες, γιατί εν τέλει οι ωφελούμενοι είναι οι πολίτες. Σίγουρα λοιπόν πρέπει να υποστηρίξουμε αυτή την κατεύθυνση. Αλλά και θα πρέπει η υπηρεσία αυτή να, γίνει, να καταστεί πιο ορατή, όπως είπα, γιατί έτσι θα μπορέσει να λειτουργήσει και καλύτερα. Εξίσου ενδιαφέρον στο σχέδιο γνωμοδότησης είναι αυτή η πρόταση ότι τα κράτη-μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να αναπτύσσουν αυτά τα κέντρα Solvit σε εθνικό επίπεδο. Και αυτό θα μας φέρει επίσης πιο κοντά στον πολίτη. Νομίζω ότι πρέπει να το υποστηρίξουμε, αλλά ε, με λίγες ακόμη τροπολογίες. Έτσι ώστε τα προβλήματα που θα έρθει να λύσει αυτή η υπηρεσία Solvit να εξακολουθούν να, τα διαχειρίζονται σε εθνικό επίπεδο. Πέραν τούτου, νομίζω ότι πρέπει να καταλήξουμε και σε έναν συμβιβασμό, όπως είπε και ο εισηγητής, για το διασυνοριακό εργασιακό δίκαιο. Και ιδιαίτερα ένα θέμα που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή είναι το θέμα της ε, προσβασιμότητας σε διασυνοριακές διαφορές. Και επειδή πιστεύουμε ότι δεν πρέπει να γίνονται καθόλου διακρίσεις, τόσο η υπηρεσία όσο και οι δικτυακοί τόποι πρέπει να είναι ανοιχτοί σε άτομα με ειδικές ανάγκες, προσβάσιμοι στα άτομα με ειδικές ανάγκες. Ε, κάτι άλλο που δεν θύχτηκε, μπορούμε πιστεύω να καταλήξουμε σε συμφωνία ως προς το Solvit και για τον τρόπο που μπορεί να βελτιωθεί έτσι ώστε να μεγιστοποιηθεί το όφελος προς όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Ευχαριστώ. Ο Φιλ Μπένιον έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ε, μιλώ εκ μέρους της Μάρια Χάρκιν. Ζητά συγγνώμη που δεν μπορεί να είναι εδώ σήμερα μαζί μας. Η Μάρια θα ήθελε να ευχαριστήσει τον εισηγητή για την καλή του δουλειά και για τις απόψεις του. Συμφωνεί με τις τροπολογίες που υπέβαλαν οι συνάδελφοι. Χαιρετίζει τις ε, τροπολογίες Μπαλτακίνο, ιδίως ε, την χρηματοδότηση και την ορατότητα και την προσβασιμότητα των δικτύων ε, Solvit, επίσης για μια πανευρωπαϊκή προσέγγιση ε, για μια καλύτερη ενημέρωση σε σχέση με τις διαδικασίες, τα, δίκτυα, τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών. Επίσης, η τροπολογία της κυρίας Παπαδοπούλου μιλά για μια συνεκτική προσέγγιση σε ολόκληρη την Ευρώπη για μια καλύτερη αναγνωρισιμότητα του Solvit. Η Μάρια συμφωνεί με όλα αυτά. Η Μάρια, επίσης μπορεί να ε, στηρίξει τις τροπολογίες για την ύπαρξη διασυνδέσεων μεταξύ του Solvit και άλλων δικτύων επίλυσης διαφορών, την τροπολογία του κ. Μπουλάνζ, επίσης για το, με τις θέσεις του εισηγητή και θα κάνει ό,τι μπορεί για να συνεργαστεί ωραία, καλά με τους εσκιώδεις εισηγητές. Ευχαριστώ πολύ. κύριε Κάστλα, θέλετε να ξαναπάρετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και για την ταχύτητα της παρουσίασης όσον αφορά τις ε, απόψεις της κυρίας Χάκιν. Θα ήθελα να τονίσω δύο ζητήματα. Συμφωνούμε όλοι για την ορατότητα. Είναι πάρα πολύ λίγοι οι πολίτες που γνωρίζουν αυτό το εργαλείο, το Solvit. Εγώ πολλές φορές το έχω πει και ως ε, συμβουλή, ε, έχω πει σε ανθρώπους χρησιμοποιήστε το και πράγματι ε, βοήθησε. Να τονίσω και κάτι ακόμη που το ξέχασα πριν, αλλά το έχω συμπεριλάβει και στην εισήγηση. Η πρωτοβουλία Solvit αυτή θα πρέπει να αποκεντρωθεί. Υπάρχει και αυτό το μοντέλο Solvit Regio, όπου προσπαθήσαμε να ε, κατατμήσουμε αυτό το, το, το, δίκτυο και σε εθνικό επίπεδο ώστε να επιτύχουμε και εγκύτητα αλλά και μεγαλύτερη ορατότητα για τους πελάτες. Ευχαριστώ λοιπόν που υποστηρίζετε και αυτό το, το, το μοντέλο Solvitregio. Ευχαριστώ. Θα εξετάσουμε στα 17 Δεκεμβρίου τις συμβαστικές τροπολογίες και θα τις ψηφίσουμε σε εκείνη τη συνεδρίαση. Ολοκληρώσαμε λοιπόν το σημείο 10 της ημέρης της διάταξης. Και περνάμε κατευθείαν στο 12, μια και το 11 παραπέμπεται στην αυριανή συνεδρίαση. Θα δώσω το λόγο στον φίλο Μπένιον που θα μας παρουσιάσει τις 22 τροπολογίες, στις συμβαστικές τροπολογίες ε, επί της γνωμοδότησής του για την οικονομική συμμετοχή των υπαλλήλων στα αποτελέσματα των επιχειρήσεων. Και θα ήθελα να αναθέσω την Προεδρία στην Αντιπρόεδρο την κυρία Σουρέτερ. Να Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είχαμε μια πρώτη συνάντηση των σκιωδών εισηγητών την περασμένη εβδομάδα και θα έχουμε άλλη μια αύριο. Θα κυκλοφορήσουμε την επικαιροποιημένη εκδοχή των συμβιβασμών απόψε το βράδυ. Δεν είμαι και σίγουρος αν είναι ήδη έτοιμο. Ε, Έλεγξα πριν από μια ώρα, αλλά δεν είδα. Ευχαριστώ τους συναδέλφους. Ήταν μια πολύ επικοδομητική πρώτη συνάντηση των σκιωδών εισηγητών. Καλύψαμε όλες τις προτινόμενες συμβαστικές λύσεις μέσα σε πολύ λίγο χρόνο και θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους και θα το δείτε αυτό και στις ε, αποδεκτές συμβιβαστικές λύσεις. Εγώ θα εστιάσω την προσοχή μου μόνο σε λίγες, γιατί στις περισσότερες καταλήξαμε με μεγάλη ευκολία στη διατύπωση. Ε, θα έλεγα. Ε, έχουμε δύο προτάσεις επαναδιατύπωσης για την ε, D και τη V από τους σοσιαλιστές και δημοκράτες με τη στήριξη των πρασίνων. Έχω ελαφρώς αλλάξει ε, την... Νομίζω ότι στην T θα πρέπει να διατηρήσουμε τη διατύπωση invites the government, «Καλή την κυβέρνηση κτλ. αν δεν έχουν αντίρρηση. Ε, οι εργαζόμενοι θα μπορούν έτσι να επιλέξουν να μην συμμετέχουν ε, στην διακυβέρνηση. Υπάρχουν και λιγοστοί άλλοι τομεί που απαιτούν περισσότερη συζήτηση. Αναμένω τα σχόλια των συναδέλφων. Τα πιο σημαντικά είναι το 19ο καθεστώ. Ε, εξ αρχή ήξερα ότι αυτό είναι δύσκολος τομέα για ορισμένα κράτη-μέλη και γι' αυτό έχω αποδυναμώσει το κείμενο αρκετά για να υπάρξει συνένεση. Καλώ τους ε, συναδέλφους να εξετάσουν τις τροποποιημένες συμβιβαστικέ λύσεις και θα το συζητήσουμε ξανά και στο μέλλον. Yeah. Επόμενη μιλήτρια είναι η Εύλην Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αρχικά να πω ότι θέλω να ευχαριστήσω βεβαίως τον εισηγητή για την πολύ επικοδομητική εργασία του. Γι' αυτόν τον λόγο και εγώ θα μπορέσω να είμαι πολύ σύντομη. Το ανέφερε. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το καθεστώς 29. Αρχικά είχαμε κοιτάξει τις ε, μελλοντικές προοπτικές με ενθουσιασμό και αισιοδοξία και δυστυχώς ε, τελικά το καθεστώς 29 γίνεται όλο και μικρότερο Πρέπει να το ξαναδούμε το ζήτημα, διότι η άποψή μου για τις ε, μέχρι στιγμής διατυπώσεις είναι ότι δεν θα πρέπει να συμφωνήσουμε με το καθεστώς 29. Προσπαθούμε να βρούμε μια διατύπωση ώστε να μην είναι εξαιρετικά αρνητική, αλλά εγώ ε, προς αυτή την κατεύθυνση θα ήθελα να πάμε. Τελευταία εβδομάδα, το είπατε κύριε Μπένιον, Έστειλα και κάποιες τροπολογίες για τα T και V. Ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας μέχρι στιγμής και είμαι πεπισμένη ότι θα μπορέσουμε να βρούμε μια κοινή λύση. Τέλος, μια παρατήρηση όσον αφορά την ε, τροπολογία από τον Σάρισα και δική μου αφορά το 24 και το 25. Εδώ μιλούμε για έναν συμβιβασμό με, πρόταση τη συγκεκριμένη διατύπωση την οποία εγώ δεν αποδέχομαι και δεν συμφωνώ διότι λέει θεωρεί ότι τα αποτελέσματα αυτά μπορούν να ενισχυθούν μέσω σταθερών θεσμών συμμετοχής των εργαζομένων. Εν... Σημειώνει ότι οι υπάλληλοι δεν έχουν απαραίτητα γνώσεις στις εκτελεστικές ε, αρμοδιότητες. Το αναφέρω αυτό διότι θέλω να τονίσω ότι δεν είναι μόνο οι, υπάλληλοι πάλι που δεν έχουν ενδεχομένως αυτές τις δεξιότητες, αλλά το ίδιο ισχύει και για τους ε, εργοδότες στην πλευρά του κεφαλαίου. Υπάρχουν ενώ, ενώ ταυτόχρονα υπάρχουν εργαζόμενοι που έχουν τέτοιου είδους δεξιότητες. Δεν θέλω δηλαδή να δημιουργηθεί ε, η εντύπωση ότι το όλο θέμα είναι οι δεξιότητες. Ε, αλλά νομίζω ότι σε αυτό το ζήτημα θα καταφέρουμε να βρούμε ένα συμβασμό. Κύριε Κάστλερ, λέει πρόεδρος, έχετε το λόγο. Ναι. Και εκ μέρου τη δικής μας ομάδας θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια. Ένα θέμα θέλω να τονίσω. Αυτή η παραπομπή στο καθεστώς 29. Δεν μπορούμε να... Δεν υπάρχει δεν υπάρχει λόγος να το αντικαταστήσουμε. Μπορούμε όμως ε, να το αναφέρουμε ως ε, δυνατότητα βέλτιστης πρακτικής. Ίσως έτσι καταφέρουμε να συμφωνήσουμε κιόλας. Να ε, θεσπίσουμε δηλαδή ένα εθελοντικό καθεστώς για εκείνες τις εταιρείες που θέλουν να το χρησιμοποιήσουν, να το αξιοποιήσουν και εκείνες που δεν θέλουν να το αξιοποιήσουν ίσως και για λόγους CSR ή διακυβέρνησης, να μην υποχρεούνται βεβαίως να το αξιοποιήσουν, αλλά να τους παρέχεται ως ένα μοντέλο, ένα πρότυπο βέλτιστης πρακτικής. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος, δεν ζητά κάποιος άλλος το λόγο, οπότε ο λόγος ξανά στον κύριο Μπενιόν. Για να τελειώσουμε αυτή τη συζήτηση. Ευχαριστώ. Ένα σχόλιο έχω μόνο προς την κυρία Ρέγνερ για την τελευταία της παρατήρηση. Όταν διαβάσετε την αναδιατύπωση θα διατυπώσετε ότι αυτό το σημείο το τροποποίησαμε για τις ε, δεξιότητες που πρέπει να έχουν οι τις γνώσεις. Και ευελπιστώ ότι θα συμφωνήσετε με τη νέα διατύπωση. Σε καμία περίπτωση θέλω να καταργήσω το καθεστώς του 29, απλώς θέλω να το αναφέρω κάπως πιο γενικά για τις ε, ε, επιχειρήσεις που θέλουν να εφαρμόσουν συντονισμό διασυνοριακό. Και το θέμα των βέλτιστων πρακτικών ούτω ή άλλως περιλαμβάνεται. Με προβληματίζει το γεγονό ότι μερικοί ε, θέλουν ε, με αναφορά του καθεστώτος του 29 να παραμερίσουμε τις βέλτιστες πρακτικές. Ελπίζω με τις τρεις ομάδες που σχολίασαν αυτό το θέμα ότι θα καταλήξουμε σε ένα αίσιο αποτέλεσμα. Ελπίζω και μέχρι αύριο γίνεται. Ελπίζουμε να... Ελπίζω πράγματι όλοι να ελπίζουμε ότι θα καταλήξουμε σε συμβουβασμό. Ναι, να πω ακόμη, έχουμε λίγο χρόνο ακόμη, διότι η ψηφοφορία για αυτό το θέμα δεν είναι ε, αύριο, αλλά στις 5 Δεκεμβρίου. Επομένως έχετε ακόμη κάποιο χρόνο για να καταλήξετε σε συμβιβασμό και μάλλον θα τεθεί στην Ολομέλεια τον Ιανουάριο ή τον Φεβρουάριο και με αυτό ολοκληρώνουμε τη συζήτηση για αυτό το θέμα. Θέμα 13, αλλά τελικά είναι το επόμενο, αλλά τελικά και αυτό αναβάλλεται για αύριο το πρωί και μάλιστα θα το συζητήσουμε ως τελευταίο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Πρόκειται για συμφωνία που είχαμε με την εισηγήτρια, ώστε να είναι αυτό το θέμα, το θέμα 13, το τελευταίο της αυριανής ημερήσιας διάταξης. Επομένως, με αυτό κηρύσω τη λήξη της συνεδρίασης και σας εύχομαι καλό βράδυ. Γεια σας.